So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs Committee. Καλό απόγευμα, Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, ε, καθυστέρησα λίγο διότι έπρεπε να καλωσορίσω του Ισραηλινούς φιλοξενούμενου ε, τον Άβι Ντίχτερ από την Κνεσέτ, που θα ε, μα μιλήσει στι 4 η ώρα. Θέμα 1 τη ημερησία διάταξη, έγκριση τη ημερησία διάταξη. είπαν παρατηρήσει όχι, άρα εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Σημείο 2, ανακοινώσει του Πρόεδρου, εγώ δεν έχω ανακοινώσει αυτή τη στιγμή. Οπότε μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών ε, της προηγούμενης συνεδρίας της 28 Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από εσά μέχρι το τέλος της συνεδρία, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Φτάνουμε στο σημείο 4 και θα ξεκινήσουμε από την επισκόπηση των διαπραγματεύσεων ε, επί τη Συμφωνία για το Θεσμικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία. Και έχουμε δύο προσκεκλημένου. Θα ήθελα να προσκαλέσω από τη μία τον κύριο Ρομπέρτο Μπαλζαρέτη, υφυπουργό και Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Και έχουμε και τον τακτικό μας ε, επισκέπτη, τον Κρίστιαν Λέφλερ, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΕΙΕΔ. Κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις ε, από μένα. Μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, ε, το, η Συμφωνία για το Θεσμικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας ε, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ε, ελπίζουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μετά την επίσκεψη του Ιούνκερ τον Νοέμβριο στην Ελβετία, ε, ενώ θα συνεχιστούν ε, ε, οι συναντήσεις εδώ στις Βρυξέλλες και οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ελπίζουμε να ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Μετά τις τεχνικές συζητήσεις, η Ελβετία θα πρέπει να έχει την συμφωνία των πολιτικών κομμάτων και του λαού σε δημοψήφισμα. Χωρίς πολλά πολλά, να δώσω πρώτα το λόγο στον Κρίστιαν Λέφνερ, και κατόπιν σε εσά κύριε Μπαλσαρέτη. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα 8 με 10 λεπτά για να έχουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εδώ και, ε, μάλλον, η τελευταία φορά που ήρθα εδώ ήταν πριν από 1,5 χρόνο με τον Ζακ Τεβαντούλ που ήταν επικεφαλή τη διαπραγματευτικής ομάδα τη Ελβετία. Αρχέ του 2017 για να σα ενημερώσουμε για το στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Ελβετία. Εκείνη την εποχή είχαμε μόλις ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, ε, λαϊκής πρωτοβουλίας κατά της μαζικής μετανάστευσης. Ε, από τότε οι σχέσεις με την Ελβετία έχουν βελτιωθεί πολύ. Όμως οι σχέσεις ακόμα δεν έχουν εδρεωθεί σε ένα σημείο ε, που θα συμβαδίζει με την πραγματικότητα ε, και τους πραγματικούς δεσμούς που μας ενώνουν. Ε, ούτε και σε σύγκριση με το δυναμικό αυτών των σχέσεων. Οπότε αυτό μπορώ να πω είναι ότι έχουμε να ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για το μέλλον. Είμαστε κοντά σε αυτό κάτι τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όμως το παράθυρο ευκαιρίας κλείνει γρήγορα. Να σας υπενθυμίσω εντάχει την σημασία των σχέσεων αυτών και για τις δύο πλευρές. Από οικονομικής πλευράς η Ελβετία είναι ο τρίτος ε, σε σημασία εμπορικός εταίρος. Ε, δεύτερος στον τομέα των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μάλιστα ένα εμπορικό πλεόνασμα, σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα. Ε, έχουμε ε, επίσης επενδυτικά συμφέροντα το 30% των επενδύσεων της Ελβετίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 4 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στην Ελβετία και 460, ε, 460.000 ε, Ελβετοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, 320.000 Ευρωπαίοι πολίτες παίρνουν τα σύνορα της Ελβετίας κάθε μέρα για να εργαστούν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τη ε, ε, ε συμμετοχή τη Ελβετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, συμμετέχει στο Σέγγεν και, το, και τη Συμφωνία ε, του Δουβλίνου για την αστυνομική συνεργασία και το άσυλο και τη μετανάστευση. Εφαρμόζει η Ελβετία το, το κεκτημένο, συμμετέχει στη Frontex, στην EU Lisa και στα συστήματα πληροφοριών όπω το SIS. Επίση, συνεισφέρει και λαμβάνει ε, κονδύλια σε αυτού του τομεί. Επίση, επίσης βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς. Εκπαίδευση, έρευνα, μεταφορές, ε, περιβαλλοντικές πολιτικές, κλιματική αλλαγή κλπ. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελβετία στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερείς οργανισμούς σχετικού με την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εφαρμογή της Ατζέντα 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ τακτικά λαμβάνει χώρα, λαμβάνει χώρα πολιτικός ε, διάλογος σε διάφορα επίπεδα, θεματικά και γεωγραφικά. Επίσης η Ελβετία συμμετέχει στις ad hoc συμφωνίες ε, σε αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σταθερότητα και την ε, διαχείριση κρίσεων όπως του κοσυφοπεδίου, το εκπαίδευση στο Μάλι κλπ δεν δεσμεύεται από τις εξω... αποφάσεις εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά ε, συνεργάζεται, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εξωτερικής δράσης. Για να εμπεδώσουμε αυτή τη σχέση χρειάζεται να συμφωνήσουμε επί ενός συνολικού ε, θεσμικού πλαισίου που θα, θα περιλαμβάνει και την συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια συμφωνία ε, θα εδραίωνε τη διμερή σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες, θα εξασφαλίσει ίσως ίδιες συνθήκες ε, από τις δύο πλευρές και μια νομική ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπόδια λόγω της έλψης μηχανισμών, κανόνων ε, για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην ε, Ελβετία. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα έδινε ρόλο στους εκπροσώπους Ελβετίας και στην συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για ένα μελλοντικό κεκτημένο. Επίσης, μηχανισμοί επίλυση διαφορών, έτσι ώστε να λύνονται ε, έντοιμα οι διαφορές μας οποτεδήποτε αυτές παρουσιάζονται. Πρόκειται για ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα στην Ελβετία. Το θέμα της συζήτησης για τους ξένους δικαστές έχει ταράξει τα νερά. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε μια πρόταση πριν μερικούς μήνες ε, η επίλυση των εφορών να ε, αναλυθεί από ε, ένα δικαστήριο, αντικειμενικό δικαστήριο τρίτων, στο οποίο όμως θα συμμετέχουν και ευρωπαϊκοί και Ελβετοί δικαστές. Σε ε, περιπτώσεις που θα χρειαστεί θα μπορούν να προσφεύγουν στο πρώτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε η ερμηνεία του δικαστηρίου αυτού να είναι ενιαία ε, ενώ το δικαστήριο αυτό, το, το, το, το, ανεξάρτητο δικαστήριο, θα έχει και περιθώριο λιγμών. Θα χρειαζόμασταν βέβαια και κοινά όργανα που θα επιτηρούν την εφαρμογή της συμφωνίας. μετά από πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων, έχουμε καταλήξει σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε προχωρήσει μάλλον σε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στο τραπέζι και χρειάζεται να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα και νομίζω ότι μπορεί να γίνει μετά από λίγες ακόμα συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Αυτό που θέλουμε δηλαδή είναι να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο κείμενο για τις κρατικές ενισχύσεις που θα ε, Προσθεθεί στην Συμφωνία Περινέρων Μεταφορών του 1999. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι δεν θα δεχτούμε συμφωνία χωρίς τέτοιου είδους διατάξεις περικρατικών ενισχύσεων. Επίσης, δεύτερον, χρειάζεται να κλείσουμε συζήτηση σε ορισμένα θέματα νομοθετικά στα οποία η Ελβετία αντιμετωπίζει πολιτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία ε, διακίνησης. Θεωρεί ε, η Ελβετία ζητά κάποια προστατευτικά μέτρα τα οποία για μας είναι υπερβολικά και θα έβλαπταν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών ε, και επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, θέλουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τι ίδιε υποχρεώσεις και να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Μέσα στο 2018 προχωρήσαμε πάρα πολύ προ μια κοινή θέση. Όχι μόνο για την επίλυση των διαφορών, αλλά και για το εύρο, το βεληνικέ της συμφωνίας, η οποία θα εμπνέεται από τη συμφωνία του 1999, αλλά και κατοπινέ κλαδικές συμφωνίε. Συμφωνήσαμε επίση ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις που βασίζονται στην Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών του 1972 αυτή τη στιγμή. Αυτή θα πρέπει να την προσαρμόσουμε στις σημερινές συνθήκες όπως οι συμφωνίες του Καναδά και της Ιαπωνίας. Αυτή η συμφωνία θα, ωφελήσει, θα ωφεληθεί και από τους μηχανισμούς της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι δυνατόν πιστεύω να κλείσουν διαπραγματεύσει, διότι πλέον έχει έρθει η ώρα να ληφθούν πολιτικέ αποφάσει. Τεχνικά είναι δυνατόν, νομικά είναι δυνατόν, εξε, ε, εξαρτώμαστε από την πολιτική βούληση. Όπω είπε και ο πρόεδρο Γιούνκερ όμω, ο χρόνο πιέζει, το τα περιθώρια στενεύουν. Ε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι, το τέλος, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, διότι αλλιώ θα επηρεαστούμε από άλλε διαπραγματεύσει που λαμβάνουν χώρα παράλληλα. Και τελειώντας να ε, σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι μία ακόμα συμφωνία, είναι μία κρίσιμη συμφωνία πλαίσιο, δεδομένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι αυτή η συμφωνία είναι προϋπόθεση προκειμένου να συμμετάσχει περαιτέρω η Ελβετία στην εσωτερική αγορά. Στόχος είναι να εδρεωθεί η διμερής προσέγγιση έτσι ώστε να μην χαθούν σταδιακά τα ωφελήματα τα οποία αντλεί η Ελβετία από τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε συμφωνίες και με άλλους εταίρους, να αναπτύξουμε νέους τομείς της εσωτερικής αγοράς, όπως η ψηφιακή εσωτερική αγορά. Το status quo θα σήμαινε ότι τα κενά στη σχέση μας θα αυξηθούν. Το ίδιο και τα εμπόδια στο μέλλον. Χρειάζεται εύρος και βάθος και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πλαίσιο για μια νομική ασφάλεια για τους φορείς που συνεργάζονται. Ε, αυτό θα βοηθήσει και τους πολίτες. Η διμερή συμφωνία, οι διμερείς συμφωνίες λειτουργούν υπέρ και των δύο πλευρών, αλλά μερικές φορές υπάρχουν τριβές και είναι απαραίτητο αυτές να λύνονται με έναν τρόπο ικανοποιητικό και προς τις δύο πλευρές. Τέλος, πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε την δυναμική συνεργασία μας, θα ανοίξουμε καινούριε ευκαιρίες και θα αντλήσουμε από αυτό το δυναμικό το οποίο κρεμεί. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Λεφνέρ. Χωρίς ε, καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην κύριο Μπαλτζάρα. Την να διαλέξτε σε ποια γλώσσα θα μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Κριστιαν Λεφλέρ για την παρουσίαση αυτή. Θα μπορούσα να είχα γράψει κι εγώ ακριβώς τα ίδια, με εξαίρεση ορισμένα σημεία, στα οποία θα ήθελα να επανέλθω. Ο Κριστιαν Λεφλέρ ε, είπε σε μεγάλο βαθμό αυτά που θα ήθελα να πω κι εγώ. Να σας δώσω τα νούμερα για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η διμερής ε, σχέση Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα νούμερα που ανέφερε ο κ. Λεφλέρ. Ε, από πλευράς Ελβετίας αυτή η σχέση υπήρχε ε, και πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, αυτό είναι βέβαιο, με κανονικές έντονες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες χώρες του πλανήτη αλλά είχαμε ακόμη μεγαλύτερε σχέσει με τι γειτονικέ χώρε. Τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία. Ε, χώρε γείτονε, ε, χώρε φιλικέ, ε, με τι οποίε διατηρούμε πολύ σημαντικέ σχέσει εδώ και αιώνε. Όπω οι οικονομικέ σχέσει που έχουμε με τη Λομβαρδία είναι εξίσου σημαντικέ με αυτέ που έχουμε με την Ιαπωνία με τη Βάδη Βιρτεμβέργη και με τη Βαβαρία έχουμε οικονομικές σχέσεις στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα μπορούσα να συνεχίσω, να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Μέσα στην ιστορία λοιπόν αναπτύξαμε μια οικονομία ε, στενά συνδεδεμένη με αυτές τις συνοριακές περιοχές. Μιλάμε όμως και τις τρεις γλώσσες πέραν αυτού ε, των γειτόνων μας. Έτσι έχουμε και πολιτιστικές, κοινωνικές σχέσεις που υπερβαίνουν την απλή οικονομία. Αυτό που συζητάμε εδώ λοιπόν είναι πώς θα διατηρήσουμε τη σχέση αυτή ως έχει, πώς θα την εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Ο Κριστιαν Λεφλέρ υπενθύμησε τις προσπάθειές μας εδώ και αρκετό καιρό για να επιτύχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στη σχέση μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα να πω ότι πριν από αυτό και μετά από την απόρριψη το Δεκέμβριο του 1992 του ΕΟΧ από την ε, Ελβετία ε, συνάψαμε καμιά εικοσαριά ε, σημαντικές διμερείς συμφωνίες που έδωσαν τη δυνατότητα στην οικονομία και στους πολίτες μας επίσης να σημειώσουν κάποια ανάπτυξη και στις δύο πλευρές των σύνορων. Τα σύνορά μας είναι ε, ανοιχτά και για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει του συστήματος Σέγγεν και του Δουβλίνου ε, έχουμε ε, αυτή τη σχέση είτε μέσω των διμερών συμφωνιών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Είναι συμφωνίες που επέτρεψαν σημαντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπήρου μεταξύ της δικής μας χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, όπως διαμορφώθηκε μέσα στα χρόνια. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να τα οργανώσουμε όλα αυτά, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις πέντε συμφωνίες πρόσβασης στην αγορά. Με στόχο να πλησιώσουμε αυτές τις ε, ε, πέντε συμφωνίες, ώστε αφενός να συνεχίσουν να λειτουργούν σωστά ή ακόμη προτιμότερα ε, καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, από τη σήμερα. Αφετέρου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε σχέσεις και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία για την πρόσβαση της Ελβετίας στην αγορά ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης. Ο Κριστιαν Λεφλέρ υπενθύμησε τα βασικά σημεία. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω δύο σημεία. Το πρώτο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Είναι σαφές ότι ευθύς εξ αρχής η Ελβετία είχε μια ιδιαίτερα επιφυλακτική θέση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Αυτό οφείλεται στη δική μας γεωγραφική θέση, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Είναι προφανές, είμαστε μια μικρή χώρα με μια πολύ ανοιχτή οικονομία μεγάλη ευκολία στις συναλλαγές, αλλά σχετικά μικρή χώρα ε, μέσα στη μέση της Ευρώπης, ανάμεσα σε πολύ μεγάλες και σημαντικές χώρες. Εμείς έχουμε ένα επίπεδο αμοιβών και κοινωνικής προστασίας επίσης πολύ αναπτυγμένο και υπέστημε τεράστια μεταναστευτική πίεση. Μεταναστευτική πίεση που ναι μεν υπήρξε πολύ επωφελής για την οικονομία μας, διότι αυτή η μεταναστευτική πίεση μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ικανότητες, ε, γνώσεις ε, ε, από τις γειτονικές χώρες, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνώσεις και ικανότητες και ανθρώπους που ίσως δεν είχαμε στις χώρες μας. Αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία λοιπόν των προσώπων την διαχειριστήκαμε αρκετά επιφυλακτικά στην Ελβετία ευθύ εξ αρχή για λόγου κατανοητού, αλλά ταυτόχρονα αυτή συνέβαλε εκπληκτικά στην ανάπτυξη τη χώρα μα. Σήμερα λοιπόν αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Αυτό το άνοιγμα της χώρας μας, αυτή την ελευθερία κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε τα μέτρα που υιοθετήσαμε για την προστασία των εργαζομένων για να αποφύγουμε το μισθολογικό και κοινωνικό dumping ώστε η αγορά εργασίας αυτή να συνεχίσει να εξελίσσεται με τρόπο που θα επιτρέπει όχι μόνο τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και το σεβασμό ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ε, ώστε να εργάζονται υπό αποδεκτές συνθήκες. Αυτό είναι ένα σημείο που συζητάμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας. Αυτό διευκολύνθηκε από την πρόσφατη οθέτηση για την, ε, της οδηγίας της απόσπασης εργαζομένων και της εφαρμοστικής οδηγίας που αποτελεί ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό το οποίο δεν θα σας κρύψω πλησιάζει στο επίπεδο που έχουμε στην Ελβετία, ε, χωρίς να θελήσω να φανώ ανακουστώ αλαζονικό. Ε, μετά, όπως είπε ο Κριστιαν Λεφλέρ, ε, αυτό που προσπαθούμε στην, στο θεσμικό πλαίσιο, στο θεσμική συμφωνία, είναι να έχουμε ένα πλαίσιο διατάξεις που να διευκρινίζουν πόσο αναγκαίο είναι και στι δύο πλευρέ των συνόρων όταν συνάπτουμε συμφωνίε να διευκρινίζονται οι, αρχ... οι αρχές, οι διαδικαστικές, η συνεργασία μεταξύ των αρχών, η διαφάνεια, σημαντικά στοιχεία, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να λειτουργήσει μια ολοκληρωμένη αγορά σωστά. Οι συγκεκριμένε διατάξει που αφορούν τι κρατικέ ενισχύσει πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτέ τι τομεικέ συμφωνίε, πιστεύω. Ε, υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, αλλά νομίζω ότι ε, είμαστε όλοι διατεθειμένοι και συμφωνούμε. Κάτι που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει μέχρι σήμερα είναι το γενικότερο περιβάλλον. Ε, ε, δεν σας κρύβω ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Δεκεμβρίου 2017 να περιορίσει κατά ένα χρόνο την αναγνώριση του ελβετικού χρηματιστηρίου έγινε δεκτή καταρχάς με έκπληξη διότι αντικειμενικά ε, πληρώνταν οι αντικειμενικές συνθήκες ε, αναγνώρισης, αλλά επίσης ε, παρενέβη ενώ η κυβέρνησή μας προσπαθούσε να επανεκκινήσει την διαδικασία για την διοργανική συμφωνία. Επίσης περιορίστηκε για ένα χρόνο αυτή η απόφαση, αλλά τώρα αμφισβητείται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λένε ότι είναι μια απτή διαδικασία και να είστε σίγουροι ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου δεν θα έχει αναγνωριστεί το ελβετικό χρηματιστήριο ως αντίστοιχο μέχρι τα τέλη του έτους. Δεν είναι πολύ ευχάριστο λοιπόν το περιβάλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές πολιτικές συνιστώσεις έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις που είναι και τεχνικές και πολιτικά σημαντικές από τη φύση τους, αλλά φυσικά αν μέχρι τα τέλη του έτους δεν δοθεί αυτή η αναγνώριση βάσει κριτηρίων ε, που δεν είναι τα αντικειμενικά κριτήρια, θα έχουμε πρόβλημα. Κάτι άλλο που μάλλον είναι καλή είδηση, η δική μας κυβέρνηση αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο μια αίτηση πίστοση 1,3 δισεκατομμυρίων για να συμβάλλει η Ελβετία στην ε, κοινωνική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1,3 δισεκατομμύρια περιλαμβάνουν ε, που περιλαμβάνουν 200 εκατομμύρια για το μεταναστευτικό σκέλος και για χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα που δεν είναι, αν είναι πλέον οι χώρες συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να συνοψίσω λοιπόν, ε, μας συμφέρει σίγουρα να διατηρήσουμε μια σχέση ε, όπως αυτή που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ε, πολύ σημαντική σχέση για την Ελβετία, όχι μόνο ουσιώδης οικονομικά, βασίζεται και στο κοινή ε, εικόνα του κόσμου που έχουμε, τις κοινέ αξίες, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τη διακυβέρνηση. Είναι μια χώρα, η Ελβετία, τόσο ευρωπαϊκή όσο και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας συμφέρει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση και να συνάψουμε μια ε, διοργανική ε, συμφωνία που θα είναι μια καλή συμφωνία που θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή τη συμβατική την νομική σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Έχουμε κάποια σημεία τα οποία ε, πρέπει να συζητήσουμε και κάποιες απαιτήσει που τα εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ από τότε που ασχολούμαι απευθεία με τη διαπραγμάτευση, δηλαδή από το Μάρτιο και μετά, έχω παρατηρήσει ότι πάντα καταφέρουμε να βρούμε μια καλή λύση σε κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται. Φυσικά τώρα πλησιάζουμε προ το τέλο των συζητήσεων αυτών Οπότε εδώ οι συζητήσει είναι πιο δύσκολε. Πάντα έτσι γίνεται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Προ το τέλο δυσκολεύουν οι συζητήσει και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα ε, πνεύμα συνεργασία, ε, αναλογιζόμενοι τα όσα μα ενώνουν αντί για τα όσα μα χωρίζουν. Και έτσι θα κλείσω. Η κατάσταση τη Ελβετία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από αυτήν άλλων χωρών. Ε, χωρών, για παράδειγμα, που θέλουν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε τελείω διαφορετική κατάσταση. Σίγουρα δεν θέλουμε διαζύγιο, αντιθέτω. θέλουμε αντιθέτως να ενισχύσουμε την εταιρική αυτή σχέση ε, που έχουμε εδώ και χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει φυσικά να υπερασπιστεί τα δικά τη συμφέροντα στο πλαίσιο αυτή τη συνεργασία και η Ελβετία επίση θέλει να υπερασπιστεί τα ελβετικά συμφέροντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you to... Ευχαριστώ και τους δύο προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστώ κύριε Παλσαρέτη που δεν έχετε σχέδια διαζυγίου. Μας απασχολεί αυτή τη στιγμή ένα άλλο διαζύγιο. Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο καταρχάς στον ε, πρόεδρο της ε, αποστολής ε, DEA, τον κύριο Γιάνν Ντόρμαν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι, όπως ακούσατε, πρόεδρος της αποστολής DEA που παρακολουθεί από κοντά τις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία. Τον Ιούλιο είχαμε την ετήσια συνάντηση με βουλευτές της Ελβετίας και Είχαμε επίσης αποστολή στην Βέρνη όπου συναντήσαμε Ελβετούς πολιτικούς. Είναι πολύ ε, κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συνάντηση με τους διαπραγματευτές τώρα που πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα σύντομα να έχουμε επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων που συνεχίστηκαν δυστυχώς για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τον Μάιο του 2014 έχουν ξεκινήσει. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, κατάλαβα ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι Ελβετοί δεν επιδεικνύουν πολύ ευελιξία όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές τους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν έχουμε εμείς κάποιο σχέδιο αναδίπλωσης, κάποιο εναλλακτικό σχέδιο και ελπίζω πραγματικά να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάνν Ντόρμαν. Τρεις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Ανδρέας Σφαπ, καταρχά. Έχουμε και τον Χέλμουτ Σόλ, σε άλλο κανεί. Ήδη έχουμε καθυστερήσει κάπω. Παρακαλώ περιοριστείτε στα δύο λεπτά ο καθένας για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τι απαντήσει. Ανδρέα Σφάπ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των διμερών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετία δεν είναι μόνο θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι και σε μεγάλο βαθμό οικονομικό θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές για τις πολύ σαφείς παρουσιάσεις τους και έχω μια σειρά ερωτήσεων. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λέφλερ. Ε, τι εκχωρήσει έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την το δικαστήριο διατησίας και αυτό δεν ξεπερνάει αυτά που είχαν σχεδιαστεί αρχικά, διότι πρόκειται για την ερμηνεία ευρωπαϊκού δικαίου και μόνο ένα δικαστήριο είναι αρμόδιο γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κύριε Λέφλερ, μήπως θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε αυτό. Ε, κύριε Μπαλσαρέτη. Η Ελβετία, εγώ γνωρίζω ότι πάντα ήταν φιλελεύθερη χώρα, είσαστε και πολύ καλοί γείτονε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο φιλελεύθερη όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων από την Ελβετία. Μήπως η Ελβετία κάνει λάθος, μήπως ως χώρα υπόδειγμα ε, της δημοκρατίας θα έπρεπε να ακολουθήσει άλλο μοντέλο, δηλαδή να έχει ε, αυστηρούς ελέγχους αλλά να είναι ανοιχτή η χώρα. Και επίσης ε, γνωρίζω από το δικό μου κρατήδιο ότι είχε απελευθερωθεί το θέμα της, των αστικών ασφαλίσεων. Στην Ελβετία λοιπόν τι γίνεται όσον αφορά τις ασφάλειες πυρός. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει σχεδιαστεί η σχετική συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ. Άννα Γκόμες, δύο λεπτά παρακαλώ. Θα ήθελα να, να ρωτήσω τον κύριο Κρίστιαν Λέφλερ, αλλά ίσως να θέλει να σχολιάσει και ο Ελβετός προσκεκλημένος μας. Οι συστάσεις του Κοινοβουλίου μας στο έγγραφο, ε, στην έκθεση για το έγγραφα του Παναμά όσον αφορά την Ελβετία σχετικά με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Οι συστάσεις του Κοινοβουλίου αυτές λοιπόν πώς ελήφθησαν υπόψη στις διαπραγματεύσεις που έχετε αυτή τη στιγμή με την Ελβετία. Διαπιστώσαμε ότι η Ελβετία είχε δεσμευτεί να καταργήσει το τραπεζικό απόρριτο, αλλά βλέπουμε ότι διατηρείται Επίσης, η φοροαποφυγή δεν είναι έγκλημα, δεν είναι αδίκημα στην Ελβετία και αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για μας. Τα διάφορα καντόνια ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές φορολόγησης, κάτι που μας ανησυχεί πολύ. Είδαμε πρόσφατα τι έγινε στη Ζηρίχη. Και όσον αφορά τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ε, όπως και η φοροποφυγή, φαίνεται να είναι τελείως εκτός ελέγχου στην Ελβετία. Υπήρξαν προσπάθειες ελέγχου από το ε, Ελβετικό Κοινοβούλιο, αλλά κάποια κόμματα τελικά ήταν κατά και τίποτα δεν επιτεύχθη. και έχουμε και το θέμα των ε, αυτών που αναφέρουν παρατυπίες, το οποίο ε, είναι επίσης πολύ σοβαρό. Όλα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας και θα πρέπει να ρυθμίζονται στη σχετική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ ο Charles Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Άννα δεν ανέφερε το περίεργο καθεστώς του Καμπιόνε Ιτάλια αλλά βέβαια η δική μου πολιτική ομάδα στηρίζει την ε, συμφωνία τη Συμφωνία Θεσμικού Πλαισίου. Εγώ όμως θέλω να ταξιδέψω στο μέλλον, τον Οκτώβριο του 2020, που μια δήλωση όπως του κυρίου Λέφλερ μπορεί να είναι αυτά που θα ακούμε από τη Βρετανία για τις μελλοντικέ τους ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί βουλευτές του κόμματός μου ισχυρίζονται ότι το, ότι το μοντέλο της Ελβετίας θα είναι η κατάλληλη λύση για τη Μεγάλη Βρετανία μετά την αποχώρησή της. Αλλά μόλις διαπιστώσουν ότι περιλαμβάνει και την ε, ε, ελεύθερη κυκλοφορία, τότε εκπλήσονται. Η κυβέρνησή σας ε, σχεδόν αγνόησε τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος, ε, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιον αξιοπρεπή συμβιβασμό. Επίσης έχετε το σύστημα όπου οι τοπικές θέσεις εργασίας μπορούν να δίδονται σε ε, ντόπιου. Ε, δυστυχώς όμως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ανακοίνωσε μέσω του Υφυπουργού ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία τέτοια δυνατότητα για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας μετά το Brexit. Το θέμα όμως είναι πώς η Ελβετία καταφέρει να πετύχει τόσο καλή διμερή συμφωνία ε, όπου να μην ε, συμπεριλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να μην έχουν συνέπειες ε, οι αποφάσεις του και να πληρώνει κατά κεφαλήν το μισό από όσα πληρώνει η Νορβηγία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε σχέση λοιπόν με την Ισλανδία και την Νορβηγία, πώς έχει καταφέρει τέτοια συμφωνία. Επίσης είναι σημαντικό το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Όσοι είναι υπέρ του Brexit ε, θα ανησυχούσαν ε, για, τις, ε, για τους κανόνες περί ενισχύσεων που επίσης ρυθμίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Από τους ελεύθερους και από τους πράσινους δεν έχουμε κανέναν. Ο κ. Σόλτς τώρα. Παρακαλώ. Τρεις επιπλέον ερωτήσεις. Αν κοιτάξει κανείς τις δημοσκοπήσεις ε, στην Ελβετία καθώς και την ε, συμπεριφορά ε, διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Ελβετίας, αναρωτιέται γιατί λένε ότι η συμφωνία πλαίσιο είναι υπερβολική. Εσείς σε τι βαθμό βλέπετε η εσωτερική συζήτηση στην Ελβετία να επιτρέψει μια μακροπρόθεσμη θεσμική συνεργασία. Μήπως ε, θα είναι περισσότερο σε στάση αναμονής η Ελβετία εσωτερικά. Άλλη ερώτηση. Η Γερμανία είναι η σημαντικότερη χώρα εξαγωγής ε, προς την ε, Ελβετία και μια τέτοια συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά τον εξοπλισμό θα επηρεάσει ε, τις εξαγωγές όπλων. Και η τρίτη ερώτηση που με απασχολεί είναι το Σαββατοκύριακο σε ελβετική εφημερίδα ε, περιγράφηκε η πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελβετία το 1991-1992, ε, καθώς και η σημερινή κατάσταση. Η συναλλαγματική ισοτιμία ε, ευρώ και ελβετικού φράγκου, το θέμα των θέσεων απασχόλησης, μήπως αποτελούν και αυτά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Okay, δεν έχουμε άλλε ερωτήσει. Εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Από ό,τι είπατε, υπάρχει ένας στόχος να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Αλλά θα χρειαστούμε άλλο ένα μήνα εδώ, οπότε πριν από το 2020 δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να επικυρωθεί η συμφωνία. Παρόλα αυτά το Συμβούλιο ε, στοχεύει στο να λάβει την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Πώ γίνεται αυτό, Δέκα λεπτά για να μα απαντήσετε. Πέντε λεπτά ο καθένα. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, Ο κ. Μπαλτσαρέτη. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, ορισμένες από αυτές ε, απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ντόρμαν, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει την ευελιξία μας όσο μπορούμε. Η κάθε πλευρά πηγαίνει στις διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες οδηγίες, διαπραγματευτικές οδηγίες και κόκκινες γραμμές. Αλλά η εντόλη που λαμβάνουμε ή λαμβάνει υπόψη και την πραγματικότητα στις χώρες μας. Το σύστημά μας ε, μας επιτρέπει να ξέρουμε αν η κοινή γνώμη είναι υπέρ ή κατά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για plan B. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο plan A και κάνουμε προσπάθειες να βρούμε μια λύση μεταξύ άλλων θεμάτων και για το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, για όλο το πακέτο. Και Πιστεύω ότι με την, νέα, την εφαρμοστική οδηγία για τις ε, αποσπάσεις εργαζομένων ε, έχουμε προσέγγιση των ε, δύο νομικών τάξεων. Και αυτό εν μέρη συνδέεται και με τα διαφορετικά νομίσματα, με την ε, αξία του ελβετικού φράγκου, με τις ιδιαιτερότητες ε, της αγοράς εργασίας της Ελβετίας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ακόμη κάποια ακόμη ε, προφυλακτικά μέτρα. Η οδηγία περί αποσπάσεων υιοθετήθηκε το 2004. Σήμερα όμως έχουμε μια νέα κατάσταση και πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτό αποτελεί σημαντική υποχρέωση για μας ε, να προστατεύσουμε τις ε, αποδοχές των εργαζομένων. Και το πώς ε, αποτελεί αντικείμενο των συζητήσεών μας. Και μία μικρή παρατήρηση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο. Πράγματι, ε, πρέπει να προσαρμοστούμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την συμφωνία. Για μας, λοιπόν, είναι δίκαιο που απορρέει από μια διεθνή σύμβαση. Συνεχίζουμε όμως να είμαστε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ε, και γι' αυτό έχουμε ειδικό δικαστήριο διατησίας ε, και όχι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ερώτηση του κυρίου Τάνοκ νομίζω απευθυνόταν προς τον Κρίστιαν Λέφλερ. Ε, στα γαλλικά τώρα. Κυρία Γκόμες, ε, οι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι συστάσεις κάθε άλλου κοινοβουλίου του κόσμου, είναι μια πηγή soft law. Τις λαμβάνουμε υπόψη. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι τις διαβάζουμε και τις γνωρίζουμε και τις λαμβάνουμε υπόψη. Ίσως από την άλλη μεριά δεν κατάλαβα καλά, αλλά η φοροδιαφυγή στην Ελβετία είναι αδίκημα. Εγώ ποτέ δεν έχω φοροδιαφύγει, αλλά θα συμβούλευα σε οποιονδήποτε να μην διαμένει στην Ελβετία και να προσπαθεί να φοροδιαφύγει, γιατί θα τιμωρηθεί. Τα καντόνια τώρα πράγματι έχουν διαφορετικά φορολογικά συστήματα, όπως και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει σχέση και με τον οικονομικό ανταγωνισμό, αλλά και με την οικονομική και φορολογική ισχύ του κάθε καντονίου. Έχουμε όμως ένα ομοσπονδιακό νόμο που καθορίζει τις βασικές αρχές όλων αυτών των συστημάτων και ένα σύστημα επιμορισμού, εσωτερικού επιμερισμού, οριζοντίως και κατακορύφως, έτσι ώστε τα λιγότερο πλούσια καντόνια να παίρνουν πόρους από τα πιο πλούσια. Υπάρχει λοιπόν μια, ένας φορολογικός ανταγωνισμός, ο οποίος όμως επανεξισορροπείται με έναν κατοπινό μεταγενέστερο επιμερισμό. Τώρα το θέμα της αναθεώρησης των νόμων για την φορολογία των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε σε αυτό ή όχι. Ε, όμως ολοκληρώνεται, η κυβέρνηση έχει εγκρίνει το νομοσχέδιο μπορεί να τεθεί σε δημοψήφισμα αν το ζητήσουν 50.000 ε, πολίτες μας και αν γίνει κάτι τέτοιο, δημοψήφισμα δηλαδή, θα γίνει το Μάιο. Μετά θα έχουμε ένα νόμο που θα είναι ένας από τους πιο σύγχρονους νόμους με όλες τις εγγύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διμερείς μας συζητήσεις προκειμένου η φορολογική ε, μεταχείριση των μεγάλων επιχειρήσεων να μην δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο φορολογούνται σωστά. Τώρα, οι καταγγέλλοντες ότι βρίσκονται σε κίνδυνο στην Ελβετία δεν το καταλαβαίνω. Άλλο οι καταγγέλλοντες όμως και άλλο τα άτομα τα οποία καταχρώνται πληροφορίες οι οποίες τους είχαν εμπιστευτεί τους, ε, όλες οι νομοθεσίες του κόσμου προβλέπουν ποινές για κάποιον ο οποίος αποκαλύπτει μυστικές πληροφορίες. Αυτό δεν αφορά καταγγελίες. Τελευταία ερώτηση. Η πολιτική συζήτηση στην Ελβετία. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε όλες τις απόψεις όλων των πολιτικών κομμάτων και σημαντικό στη συζήτηση αυτή είναι εάν αφήσουμε κατά μέρος την προέλευση κάποιων πολιτικών ιδεών και εξετάσουμε το περιεχόμενο, Αυτή είναι η τέχνη επίτευξης μιας συμφωνίας για να πετύχουμε την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Γνωρίζουμε ότι κάποια πολιτικά κόμματα είναι κατά της προσέγγισης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς εξετάζουμε το περιεχόμενο. Οι εξοπλισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την ε, Συμφωνία Θεσμικού Πλαισίου. Η ερώτηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με την αγορά εργασίας. Ναι, πράγματι η αγορά εργασίας ε, της Ελβετίας ε, έχει γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, επειδή και η συναλλαγματική ισοτιμία είναι τόσο ευνοϊκή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λέφλερ. Um, um, Ευχαριστώ. Που εν συντομία αν έκανε πολλές παραχωρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς δεν το πιστεύω, αλλιώς δεν θα τις είχα κάνει. Πιστεύω ότι ειδικά όσον αφορά το δικαστήριο το σημαντικό ζήτημα εδώ ήταν να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση που να σέβεται την ε, αυτονομία της ελβετικής νομικής τάξης ως αξιόπιστο εταίρου ε, μη ε, κοινοτικού και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως του ανώτατου δίδυτη όσον αφορά την νομοθεσία που αφορά την εσωτερική αγορά. Πιστεύουμε εμείς αυτό το συνδυασμό ενός συστήματος επίλυσης διαφορών και οτιδήποτε σχετίζεται με ευρωπαϊκή νομοθεσία το παραπέμπουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια υποχρεωτική προκατακτική απόφαση και αυτό αποδεικνύει την προσέγγιση μας. Τώρα τα χρονοδιαγράμματα, το εναλλακτικό σχέδιο του Plan B, δεν έχουμε Plan B, ούτε μελετάμε Plan B, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμη το Plan A, το πρώτο σχέδιο. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να το κλείσουμε στο χρονοδιάγραμμα παρότι είναι στενό αλλά θέλουμε να το τηρήσουμε. Κάποια ζητήματα είναι δύσκολα. Αναφέρθηκαν κάποιε κόκκινε γραμμέ. Ένα από τα λίγα καλά πράγματα που έχουμε αποκομίσει από αυτέ τι διαπραγματεύσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Ε, ξέρετε, με τον καιρό τα χρώματα χάνουν τη λάμψη τους και οι κόκκινες γραμμές γίνονται λιγότερο έντονες. Ε, πιστεύουμε ότι αν κλείσουμε τώρα, σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει κάποιο συμφέρον ε, παρά τις ε, μακροχρόνιες διαδικασίες για την κύρωση των κρατών μελών και την ελβετική διαδικασία κύρωσης. Αν λοιπόν επιτύχουμε συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντό ε, τη παρούσα θητεία, αυτό θα μα βοηθούσε. Αυτό θα στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα για τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ δεν πάω να είμαι αισιόδοξο. Αυτό επιθυμώ εγώ. Το ζήτημα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής είναι σημαντικό. Εργαζόμαστε στενά, συνεργαζόμαστε με την Ελβετία γι' αυτό. Θέλαμε η Ελβετία να ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φορολογικές δομές ε, και οι φορολογικές αρχές ε, να θεωρούνται συνεργατικές φορολογικές αρχές. Ε, υπήρξε ένα δημοψήφισμα στο ενδιάμεσο. Όλοι θα πρέπει να σεβαστούμε προφανώς την έκφραση της, της ε, λαϊκής βούλησης. Έχουν γίνει κάποιες ε, προσαρμογές και όπως είπε και ο Ρόμπερτο Μπαλσαρέτη, ελπίζουμε ότι μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι θα έχουμε την πλήρη σύγκληση και τη συνέχιση της συνεργασίας σας στον πολύ σημαντικό αυτό τομέα. φοβούνται κάποιοι ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου στην Ελβετία, αλλά ουσιαστικά ελάχιστα είναι εκτός ελέγχου. Πολλοί κόσμος όμως φοβάται ότι συμβαίνει το αντίστροφο. Το ταξίδι στο χρόνο του Charles Τάνοκ, ε, δύο χρόνια από τώρα, στο 2020, μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου τώρα και όπως υποθέτουμε σε δύο χρόνια, ε, δεν πάει να είναι τελείως διαφορετική από την Ελβετική. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να σταματήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτήν, ούτε να δεσμεύεται από του κανόνε τη εσωτερική αγορά. Η Ελβετία θέλει να διατηρήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, των ανθρώπων και θέλει να συμμετέχει και σε άλλα ε, τμήματα τη ε, ενιαία αγορά και να δεσμεύεται από του κανόνε. Αν αυτό επιθυμούσε και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ω μοντέλο την Ελβετική Συμφωνία. Αλλά δεν βρισκόμαστε σε τέτοιο στάδιο σήμερα. Συνεπώ, οι διαπραγματεύσει διαφέρουν σημαντικά. Και θα πρέπει να εξεταστούν βάσει ξεχωριστών κριτηρίων. Η συμβολή τη Ελβετία ε, στο Ταμείο Συνοχή είναι λιγότερο από το μισό από τη συμβολή τη ε, Νορβηγία, αλλά δεν συμμετέχει σε ολόκληρη την ενιαία αγορά η Ελβετία όπω η Νορβηγία, οπότε αναλογικά θα συμμετέχει στο Ταμείο Συνοχή ευρέω και συμφωνώ με τον ε, κύριο Μπαλσαρέτη. Πιστεύω ότι το θέμα της παραγωγής και εξαγωγής όπλων δεν αποτελεί κομμάτι των διαπραγματεύσεων μια συμφωνία πλαίσιο και τονίζω η συμφωνία πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό που, που ονομάζεται. Ε, δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας σε ουσιώδεις τομέα ανατομέα, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο πλαίσιο πιο σαφές, πιο προβλέψιμο με ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους εταίρους Ελβετούς και Ευρωπαίους. Εξίσου, ανοίγοντας δυνατότητας, ενδυναμώνοντας τους συμμετέχοντας και επιτρέποντάς μας, ελπίζουμε να εξελίξουμε περαιτέρω τη σχέση μας και να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο. Ήταν πολύ υποφελή αυτή η ανταλλαγή απόψεων στην ΑΦΕΤ και καλή τύχη για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων αύριο. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμά στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί σα για να βελτιώσουμε τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία. Καλή σα τύχη. Και ευχαριστώ και του συναδέλφου από την Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετία που βρέθηκαν εδώ. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Ήδη έχουμε 20 λεπτά καθυστέρηση. Φάμπιο Καστάλντο, ε, σε εσά βασιζόμαστε να δράσετε γρήγορα. Διότι ε, οι Ισραηλοί μα προσκεκλημένοι περιμένουν. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Για, σε αυτή την πρώτη ανάγνωση του δικού σας σχεδίου γνωμοδότησης ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την Ευρωπαϊκή Δεφική Εργασία. Μπορείτε, ναι, μπορώ. μπορώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω γνωρίζετε, το θέμα αυτό εντάσσεται στι ε, συζητήσει που σχετίζονται με το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για τον κανονισμό για τα νέα προγράμματα εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη. Ονομάζεται Interreg. Η συμμετοχή τη Επιτροπή μα Πρόεδρος, μπορώ να παρακαλέσω όλους όσοι σκοπεύουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα να αποχωρήσουν χωρίς φασαρία και δυνατές συζητήσεις και διαπληκτισμούς. Είναι δυνατόν αυτό μεταξύ ενηλίκων. Ευχαριστώ. Όπως σας έλεγα συνάδελφοι, εντάστε αυτό το αρχείο στις συζητήσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον κορονισμό για τα νέα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Ονομάζεται Interreg. Η συμμετοχή της Επιτροπής μας εξηγείται από το γεγονός ότι τα προγράμματα Interreg μπορούν να ενδιαφέρουν και τις χώρες ε, ε, προς προσχώρηση της γειτονίας ε, αλλά και τη Ρωσία, την Ελβετία, το Μονακό. Γι' αυτό οι σχέσεις με τα ΕΠΑ και NDICI θα βοηθήσουν και το Interreg και είναι σημαντικοί παράγοντες για αυτόν τον κανονισμό. Η πρόταση της Κομισιόν έχει κάποια καινοτόμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τον επανακαθορισμό των στοιχείων συνεργασίας με τη δημιουργία δύο νέων στοιχείων, το 3 για τις ε, εξόχως απομακρυσμένες ε, περιοχές και την 5 για τις περιφερειακές επενδύσεις σε θέματα καινοτομία και η διασυνοριακή διάσταση που θα επικεντρώνεται κυρίως ε, στα εσχερσαίες σχέσεις ε, όπου θα ενταχθούν ε, και οι θαλάσσιες ε, σχέσεις και παραμεθόρειες περιοχές. Αυτό με πείθει λιγότερο, γι' αυτό έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες για να επανεντάξουμε τη θαλάσσια συνεργασία στη διασυνοριακή συνιστόσα του κανονισμού συνεχίζοντας ε, τη σημερινή ε, περίοδο προγραμματισμού 14 με 20. Έχουμε τα ή ε, πολλά θαλάσσια όρια, σύνορα, ειδικότερα στην Νότια Ευρώπη και είναι κρίσιμη σημασία. Η πρόταση αλλαγή που κάνει η Κομισιόν θα θέσει σε κίνδυνο τα προγράμματα που θα προσέθεταν αξία όπως Ιταλίας, την Ισίας για παράδειγμα, αλλά θα ε, δυσκόλευε προγράμματα διασυνοριακά με εταιρικέ χώρε ε, σε εποχέ που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε στενότερε σχέσει με τι χώρε στην άλλη πλευρά τη Μεσογείου. Με αμοιβαία συνεργασία για αμοιβαία ωφέλη. Ένα δεύτερο νέο στοιχείο είναι η ένταξη τη ε, προγραμμάτων εξωτερική συνεργασία στην Interreg. Από τη μία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απλούστευση των διαδικασιών, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες έχουν ιδιαιτερότητες ε, στρατηγικές ε, και γι' αυτό μέσω τροπολογιών προσπαθώ να κάνω δύο πράγματα αφενός ε, να αναφέρονται οι κανονισμοί ΙΠΑΤΡΕ και NDICI και τα προγράμματα Interreg να συμπληρώνουν αυτά τα όργανα που υπάρχουν ήδη, οι πιστώσεις, οι στόχοι και οι αρχέ θα πρέπει να αναφέρονται στου αυτού του κανονισμού. Και επίση αλλάζω ορισμένα χρονοδιαγράμματα. Όταν αυτέ οι τρίτε χώρε συμμετέχουν σε προγράμματα Interreg, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα διοικητικά του συστήματα δεν είναι τόσο ρεπτυγμένα όσο τα δικά μα και δεν ακολουθούν του ίδιου κανόνε. Οπότε μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Οι υπόλοιπε τροπολογίε αφορούν μικρέ τεχνικέ προσαρμογέ και δεν αλλάζουν την ουσία του κανονισμού. Συνάδελφοι, το Ιντερέγκ έχει παίξει ρόλο κλειδί τα τελευταία χρόνια στην προσέγγιση των λαών τη Ευρώπη και πέραν τη Ευρώπη. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα είναι 10 δισεκατομμύρια. Ε, ε, έχει μειωθεί από 10 δισεκατομμύρια σε λίγο παραπάνω από 8. Οπότε πρέπει να κάνουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων ώστε να υπάρχει προσθέμενη αξία από τα προγράμματα. Και είμαι βέβαιο ότι μαζί με του κοιόδη θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε ε, παρκώς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ όλου σα. Ευχαριστούμε Φάμπιο Καστάλντο. Τέσσερα λεπτά μιλήσατε. Μπράβο. Τρία γιατί με σταματήσατε. Από τους Κιώδης λοιπόν ο κύριος Αντάμοφ του Έλκο, ο κύριος Πάσκοφο από τους σοσιαλιστές Σούλτς από την ΚΟΕ. Ξέχασα κάποιον. Οι τρεις σας λοιπόν έχετε δύο λεπτά ο καθένας κύριε Αντάμοφ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Σουίτσα γιατί δεν κατάφερε να είναι εδώ σήμερα. Ως και ό,τι συγγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καστάλτο. Γνωρίζει τις ε, τροπολογίες που προτείνει ο κύριος Καστάλτο και έχει τις εξής προτάσεις. Η κυρία Σουίτσα θέλει να αναγνωριστεί η θέση του εισηγητή ότι ο το σχέδιο κανονισμού Interreg ήδη προβλέπει ότι ποια ποσά από τους χρηματοδοτικούς φακέλους της, του μέσου γειτονία και του μέσου προενταξιακής βοήθειας θα αφιερωθούν στο Interreg. Χρειαζόμαστε μια ευελιξία. Από την άλλη μεριά, η σκιώση γητρία προτείνει να συμπεριληφθούν στο Interreg και τα προγράμματα διασυνορικής συνεργασίας για θέματα ναυτιλίας. Όμως ο κ. Καστάλτο έχει μια διαφορετική προσέγγιση από αυτήν του εισηγητή της Ρέτζη. Θα ήθελα να ρωτήσει τον κύριο Καστάλτο γιατί έχει ε, αντικαταστήσει τη λέξη adjacent με το maritime στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Πάσκο. Μιλώ εκ μέρους του συναδέλφου Πιτσούλα, ε, που προφανώς βρίσκεται στην διακατάσταση με την κυρία Σουίτσα. Έχει προβλήματα στην άφηξη, μια και έρχονται από την ίδια χώρα. Ο κ. Πιτσούλα χαιρετίζει την ε, ε, συνεργασία, την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και θεωρεί ότι ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Λέει όμως επίσης ότι σήμερα η, ο ευρωσκεπτικισμός και η, ε, οι εθνικισμοί μειώνουν την ε, αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αυτής. Αρχικά οι ανησυχίες ήταν κοινωνικονομικέ. Πιο πρόσφατα οι ανησυχίες που εκφράζονται έχουν σχέση με την μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια. Ο κ. Πίτσουλα καλωσορίζει τους κανόνες αυτούς που είναι λιγότεροι και πιο σαφείς, προκύπτουν από το νέο σύστημα διαχείρισης και αναφέρει την δυνατότητα να ενισχυθεί η συνεργασία στην Μεσόγειο ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Thank you, Jan Und nun Scholz, bitte. Και τώρα ο Χέλμουτ Σόλτ, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσέγγιση του, αλλά θα ήθελα να εκφράσω και μία άποψη που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντική όσον αφορά τα ε, προγράμματα Interreg συγκεκριμένα μέτρα που στο παρελθόν δρομολογήθηκαν και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή τους, πώς θα συνεχιστούν στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρξει διακοπή κάποιων προγραμμάτων. Και γενικά οι πόροι αυτοί πώς θα διατεθούν σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε, το Συμβούλιο προβλέπει μείωση και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα προγράμματα του Νότου, αλλά και τα προγράμματα που έχουμε στη Γερμανία, για παράδειγμα στα σύνορα με την Πολωνία ή τα σύνορα με την Τσεχία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπάρξει μείωση των πόρων και να υπάρξει συνέχιση των προγραμμάτων αυτών, διότι αποτελούν σημαντικό μέσο στα κράτη-μέλη και στις διασυνοριακές περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλμουντ Σόλς. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Φάμπιο, θέλεις ε, να κάνεις κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Γενικά έχουμε μία συνένεση πιστεύω και εκτίμηση άκουσα για τις προσπαθίες μου να αναφερθώ εν συντομία στα όσα υπόθηκαν από, τους, από τον συνάδελφο που αντικαθιστά την ε, κυρία Σουίτσα, τον συνάδελφο από το ΕΛΚ. Αντιλαμβάνομαι ότι γενικά ε, υποστηρίζεται τη βάση. Ίσως η συναδελφός να βλέπει κάποιο πρόβλημα ε, για τη λέξη adjacent. Εγώ να συζητήσω με τη συνάδελφο αν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναφέρεται αυτή η λέξη το γειτονική γιατί διακυβεύονται σημαντικές πολιτικές πτυχές να βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Αντιπρόεδρου Πάσκου εξ ονόματος του κυρίου Πίτσουλα από ό,τι κατάλαβα, κατάλαβα το πνεύμα των προτάσεων και ειδικότερα το πρόβλημα της μετανάστευσης, της ενίσχυσης της μεσογειακής συνεργασίας και σε αυτό μπορούμε να βρούμε σημεία συνεννόησης, δεδομένου ότι το ίδιο θέμα ανησυχεί και εμένα. Και τέλος, ο συνάδελφος Σόλτς αναφέρθηκε στις περικοπές, αλλά δεν θέλησαμε εμείς τις περικοπές. Η Κομισιόν τις επέβαλε και μπορεί να κάνει και άλλες το Συμβούλιο. Οπότε εμεί ως Κοινοβούλιο πρέπει να το επερασπιστούμε τον προπολογισμό του προγράμματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό δεδομένου το πόσο σημαντικό είναι. Ε, και για θε... Οπότε εκεί έχουμε σύγκληση απόψεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φάμπιο Καστάλντο. Συνάδελφοι, ευχαριστώ για τα σχόλια. 15 Οκτωβρίου, 11 η ώρα το πρωί είναι η προθεσμία τροπολογιών και 21 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ΑΦΕΤ. Έχουμε κάποια καθυστέρηση 15 ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε αμέσως στο σημείο 6. Ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ΚΝΕΣΕΤ. Ανταλλαγή απόψεων που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Και ε, καλωσορίζω και τα δικά της μέλη. Αγαπητοί συναδέλφοι, με μεγάλη μας τιμή καλωσορίζουμε τον κύριο Άβη Ντίχτερ, Πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα τη ΚΝΕΣΕΤ. Καλώ ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ καθίστε. Και οι συναδελφοί από την αντιπροσωπεία ε, των σχέσεων με το Ισραήλ ε, το 2017. Θα θυμάστε πόσο ωραία μας φιλοξένησαν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Έχουμε άλλα δύο μέλη της Κνεσέτ που θα ήθελα να καλωσορίσω. Ε, σταθείτε όρθιες, παρακαλώ, η κυρία Ανατβέρκου από το κόμμα Λιγκούντ. Καλωσορίσατε η κυρία Ρόζιν από το Έξπαρτη ε, και Σαλόμ Έχουμε τους φίλους εδώ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Κνέσετ ε, με την Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Έχουμε καλή σχέση εδώ και χρόνια για σημαντικά ζητήματα, ειδικότερα για θέματα ασφάλειας και σταθερότητα στην περιοχή και φυσικά για την ειρηνευτική διαδικασία ή ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Ντίχτερ είναι ο λόγος για τον οποίο τον καλέσαμε εδώ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για να συζητήσουμε την ε, Ισραηλινή οπτική γωνία για τις ε, σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα την κατάσταση στη Συρία και το ρόλο της Ρωσίας και του Ιράν εκεί. Όπως επίσης και τη σταθερότητα στο Λίβανο και την ασφάλεια εκεί πολλά ζητήματα σημαντικά εδώ της Επιτροπής μας, είναι σημαντικά και για τη δική σας χώρα. Σας δίνω κύριε Πρόεδρε Ντίχτερ το λόγο και θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μακάλιστερ, πέρσι όταν η Επιτροπή σας ήρθε στο Ισραήλ και σας φιλοξενήσαμε, συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συνήθως μιλούμε για τις ε, γειτονικές χώρες ως ε, εχθρούς. Όμως τα μαθηματικά στη Μέση Ανατολή λειτουργούν προφανώς διαφορετικά. Συρία, Αίγυπτος και Ιορδανία, τρεις αραβικές χώρες. Ε, γειτονικές έχουμε συνθήκη ειρήνης με την Αίγυπτο και την Ιορδανία και τώρα έχουμε τέσσερις, τέσσερα εχθρικά κράτη. Πώς έγινε αυτό. Έχουμε το Λίβανο που εξαιτίας της Χεσμολά έχει γίνει εχθρικό κράτος. Δεν σε, ε, χρωστώ κανένα σεβασμό στην Χεσμολά, αλλά δυστυχώς ε, ε, ενώ σε 19 χώρες ε, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται προσπάθεια να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεσμολάχ. Ε, είμαι πολιτικός εδώ και 47 χρόνια. Μεταξύ των μουσουλμανικών τρομοκρατικών ενώσεων ποτέ δεν έχω δει καμία περίπτωση όπου να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην στρατιωτική πτέρυγα και την πτέρυγα ασφάλειας. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να βρείτε παραλυσμούς ανάμεσα στον ΕΤΑ και τον Πατασούνα, τον, ε, τον, Ήρα και τον Σινφέιν κλπ. Αλλά στη Μέση Ανατολή αυτά, αυτές οι διαχωρισμοί δεν λειτουργούν. Τα τελευταία 25 χρόνια δημιουργήθηκε ένα τρομοκρατικό κράτος μια τρομοκρατική οργάνωση, κυρίως όμως την τελευταία δεκαετία, που ε, απειλεί την ισορροπία. Το Ιράν λειτουργεί με δύο αντιπροσώπων. Έχει πέντε αντιπροσώπους. Ό, σχεδόν όλοι είναι αντιμάχονται τον Ισραήλ. Εσμπολάχ, η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ, κυρίως στη ροίδα, τη της Γάζας, η πολιτοφυλακή των Σιτών στη Συρία προκειμένου να παίξει ένα τρομοκρατικό ρόλο ε, μέρος της Συρίας εναντίον του Ισραήλ και η Χούτι στην Ιεμένη που κάθε εβδομάδα στέλνουν, εκτοξεύουν Ιρανικούς πυράβλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Όταν προσπαθούμε να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι το Ιράν. Το Ιράν προσπαθεί να στείλει ε, ε, μέσω της Συρίας στο Λίβανο πυράβλους ακριβίας ή μέσα εκτόξευσης πυράβλων και προμαχικών ακριβίας. Αν είχα έρθει εδώ πριν από 7 χρόνια, ενδεχομένω θα είχα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, μιλώντα για, για το Παλαιστινιακό. Όμω τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης έχει γίνει τρίτη τέταρτη σε σημασία στην περιοχή μας. Όχι πως λύθηκε. Αλλά ενώ, όσο μιλάμε για της λύσης του ενός των δύο κρατών, ε, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε μια λύση τριών κρατών. Γιατί έχουμε την Χαμάς, η οποία έχει ανεξαρτοποιηθεί μαζί με τους μουσουλμάνους αδελφούς που υποστηρίζονται και έχουν δημιουργήσει ένα κράτος εν κράτη. Και την τελευταία επίσκεψη του κυρίου του κυρίου ε, Αμπάση, η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Αμπά στην ε, Λωρίδα τη Γάζα ήταν πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Πώ είναι δυνατόν ο πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή να μην μπορεί για 10-11 χρόνια να επισκεφτεί τη Λωρίδα τη Γάζα. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια τρομοκρατική οργάνωση Χαμά που διοικεί την Λωρίδα τη Γάζα τα τελευταία 10 χρόνια ε, μετά τον, το παραξικόπημα που έγινε εκεί. Αλλά να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω Πόσοι από εσά αντιλαμβάνονται ότι προκειμένου κανείς να γίνει υπάλληλο της Παλαιστινικής Αρχής έχει δύο αναγκαίες λύσεις. Ο πρώτη, η πρώτη λύση, ο πρώτος τρόπος είναι να κάνει αίτηση. Ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ πιο ασφαλής να κάνει μια τρομοκρατική επίθεση, να συλληφθεί από το Ισραήλ ή να σκοτωθεί από το στρατό. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να γίνει κανεί πάλι, στην στην αρχή. Χτε, για παράδειγμα, ένα τρομοκράτη. Στη δυτική όχθη άνοιξε πυρ εναντίον εργαζομένων μια βιομηχανίας, ενό εργοστασίου και σκότωσε δύο από αυτού, δύο Ισραηλινούς. Μια νεαρή γυναίκα που είχε και ένα παιδί και έναν άλλο άντρα που είχε τρία παιδιά και τραυμάτισε και ένα τρίτο. Ο τρομοκράτης θα συλληφθεί. Διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά θα συλληφθεί. Ζωντανός ή νεκρός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ξέρει πολύ ζωντανό είναι Παλαιστινική Αρχή χτες εγινε υπαλληλο της παλαιστινικη ένα νόμο που λέει ότι αν φυλακιστεί στο Ισραήλ λαμβάνει έναν μηνιαίο μισθό. Αν μάλιστα καταδικαστείς για περισσότερο από 13 χρόνια, λαμβάνεις ένα μισθό περίπου 3.500 δολαρίων το μήνα. Εκ του νόμου. Η Παλαιστινιακή Αρχή αμείβει κάθε χρόνο με ένα συνολικό ποσό 400 εκατομμυρίων δολαρίων τους τρομοκράτες. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε με τρομοκράτες που έχουν δράσει στην Ευρώπη. 400, εκατομμύρια δολάρια το χρόνο πηγαίνει σε αμοιβέ τέτοιων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα το οποίο μιλάει για ειρήνη, για καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ε, η στήριξη αυτού του καθεστώτος προς την τρομοκρατία είναι κάτι που πρέπει να το σταματήσουμε. Εμείς πριν από μερικούς μήνες περάσαμε ένα νόμο που λέει πώς σκοπεύουμε να σταματήσουμε αυτή την επίσημη χορηγία της τρομοκρατίας εκ μέρους της Παλαιστινικής Αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Δίχτερ, για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Έχουμε 25 λεπτά το πολύ για μια ανταλλαγή απόψεων τώρα. Έχουμε πολλά αιτήματα από πολλούς ομιλητές. Να δούμε λίγο τον κατάλογο, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε και τον χρόνο. So, I have request to speak from... Έχει ζητήσει να μιλήσει η κυρία Γκόμες, ο κύριος Καρν, ο κύριος Μπέλντερ, ο κύριος Φανόρδεν, η κυρία Φωτίγκα, ο κύριος Βάγκελ, ο κύριος Μπούχνερ, ο κύριος Κάουσον ο κ. Αστροβίσιος, κάποιος άλλος. Εννέα έχουν ζητήσει λοιπόν το λόγο. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του προσκεκλημένου μας. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είναι τιμή σας που υποδεχόμαστε εδώ τον κύριο Ντίχτερ. Εγώ όχι, εγώ είμαι διασμένη και θέλω να το πω σαφώς μπροστά στον κύριο Ντίχτερ γνωρίζοντας ότι υπήρξε επικεφάλης ε, της Ισραηλινής Συνπέντ ε, που υπονόμευσε με την πολιτική του τη σχέση με την Παλαιστίνη με στοχευμένες δολοφονίες πολλοί κόσμος ε, σκοτώθηκε σε διάφορες δολοφονίες στη Γάζα από το 2001 κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου ακόμη και από την Αμερική και υπήρχε και η πιθανότητα να συλληφθεί για εγκλήματα πολέμου το 2007 ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ο πρώτος νομοθέτης που ε, ξεκίνησε το ρατσιστικό σκέλος του κράτους του ε, καθορίζοντας ως δεύτερης κατηγορίας πολίτες τους ανθρώπους, τους πολίτες του κράτους του που είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Εγώ είμαι μέλος εδώ του κοινοβουλίου μας, είμαι διπλωμάτης και συζητώ με όλους και με το διάβολο ακόμα, αλλά θέλω να πω δεν έχω καμία ερώτηση προς τον κύριο Ντίχτερ. Όσα είπε είναι, ε, είναι, είναι πολεμοκάπηλος. Και κάνει ε, οτιδήποτε άλλο παρά να βοηθά να επιληθεί με μια Λύση δύο κρατών αυτό το πρόβλημα μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Δεν θέλω να κάνω καμία ερώτηση, απλά ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άννα Γκόμες. Πιστεύω να καλό θα ήταν να ακόμη και αν δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις με τους συναδέλφους μας από Ευγένεια να πρέπει να πούμε ότι είμαστε ε, είναι τιμή μας που έχουμε εδώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ενός ξένου κοινοβουλίου. Πάντα είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε μέλη οποιοδήποτε κοινοβουλίου όπως γνωρίζετε. Ο κύριος Πέτρε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης. Διαλύθηκαν οι οικογένειες λόγω αυτού, ε, αλλά θα ήθελα να πω στον κύριο Ντίχτερ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι σχέσεις της, ε, ε, του Κοινοβουλίου μας με την ΚΝΕΣΕΤ και έχω μια ερώτηση η Επιτροπή σας Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας ε, τι θα κάνει για να ενισχύσει τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ και επίσης ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και την Κνέσετ και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτήν. Λυπάμαι που η προλαλή σας, ε, μίλησε έτσι. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό σας, κυρία Κομές. Πώς βλέπετε επίσης ε, τις, μελλοντικέ ε, μελλοντικές επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Με την κυρία Μογκερίνη εργαζόμαστε με στόχο μια λύση με δύο κράτη. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ο Ιβο Βάγκλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ναι, θα μιλήσω τη μητρική μου. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Είχα και εγώ αντίστοιχη θέση με τη δική σας στο Κοινοβούλιο της Σλοβενίας. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ε, το κεντρικό μήνυμα της εισαγωγής σας, δηλαδή η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ είναι κάτι που θέλουμε όλοι μας. Θέλουμε το Ισραήλ να είναι ασφαλές, να μην υπάρχουν επιθέσεις, να μην υπάρχουν απειλές τρομοκρατίας. Θα θέλαμε η νέα γενιά σας ε, να ζει ευτυχισμένη σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Ωστόσο, ε, άκουσα και εγώ τις πληροφορίες που ανέφερε η κυρία Γκόμες και θα ήθελα να συμμεριστώ τις ανησυχίες της. Επίσης, αναρωτιέμαι τι θα απομείνει εάν ε, νιώθουμε οργή και έχουμε επιθετικές διαθέσεις. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε λαμπρή σταδιοδρομία και ότι κατήχατε υψηλές θέσεις και είχατε πολύ δύσκολα καθήκοντα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην πολιτική και στη διπλωματία υπάρχει μια μαγική λέξη, ο διάλογος, που βοηθάει να επιλύσουμε προβλήματα. ο διάλογος απουσιάζει στη σχέση Ισραήλ και Παλαιστίνης. Και δεν με πείσατε σήμερα ότι πράγματι ε, θέλετε τον διάλογο με την Παλαιστίνη. Ευχαριστώ κύριος Πούχνερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Frage, was die zu dem Iran beziehungsweise... Έχω μια ερώτηση σχετικά με το Ιράν και την ε, συμφωνία για πάυση των ε, ενεργειών ε, εμπλουτισμού του ουρανίου από πλευράς του Ιράν. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που είναι κατά της συνέχισης της συμφωνίας αυτής. Ειδικά το Ισραήλ, ειδικά για το Ισραήλ διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες πάυση των δραστηριοτήτων αυτών από πλευρά του Ιράν. Εάν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και τα άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής ε, θέλουν τέτοια όπλα, εάν βομβαρδιστούν οι, ε, εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, τι θα γίνει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ, Ιγκούε. Κ. Κόσο. Δεν πρόκειται να θέσω κάποιο ερώτημα στον προσκεκλημένο σας. Γιατί οι μόνε ερωτήσει που θα ήθελα να απαντήσει ένα εγκληματίας πολέμου είναι οι ερωτήσει του εισαγγελέα, ε, του δικαστή, του ανακριτή ή του, ε, των δικηγόρων. Πρόκειται για έναν εγκληματία πολέμου ο οποίος ε, στήριξε βασανιστήρια εναντίον Παλαιστινίων συλληφθέντων και διέταξε ε, δολοφονία όχι μόνο ε, ανθρώπων της Χαμάς αλλά και πολλών αμάχων μεταξύ αυτών παιδιών και γυναικών. Είναι μάλιστα ένας από αυτούς που πρόθεσαν τον καινούριο νόμο για το κράτο έθνος, κράτος έθνος ε, του Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν μαζί όπως επίσης και η διάκριση μεταξύ ε, Ισραηλινών και Αράβων δεν έχουν καμία σχέση με τις ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να καταγγείλουμε την εταιρική σχέση με το Ισραήλ, γιατί την παραβαίνει το Ισραήλ. Εσείς πρόεδρε θα όμως, θα έπρεπε επίσης να ξέρετε και να θυμάστε ότι η κυβέρνηση του ανθρώπου έχετε δίπλα σας μας απαγορεύει, απαγορεύει σε εμάς τους ευρωβουλευτές και τις Ευρωβουλευτίνες από το 2011 και μετά να μπούμε στην Γάζα. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος μας το απαγορεύει και εμείς τους τρώνουμε το κόκκινο χαλί. Δεν θέλω να βρίσκομαι καν στον ίδιο χώρο με έναν εγκληματία πολέμου και φεύγω γιατί έχω αειδιάσει. Ο κύριος Uh, thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε κοινοβούλιο με 753 μέλη και θα ήθελα να ε, διαβεβαιώσω τον κύριο Ντίχτερ ότι έχει πολλούς φίλους εδώ στο κοινοβούλιο και ότι τον καλωσορίζουμε. Είναι άνθρωπος ε, με λαμπρό παρελθόν, είναι ευγενής και ε, καταπολεμεί εδώ και πολλά χρόνια την τρομοκρατία. Γι' αυτό σας καλωσορίζουμε εδώ. Θα ήθελα να αποστασιοποιηθώ από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε από συναδέρφους της αριστεράς, που ε, έχουν αιμονή στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό δεν βλέπουν ε, τις πραγματικές συνθήκες σε ένα μέρος του κόσμου όπου υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Εγώ θα διαφωνούσα στο ότι Κάνετε διάκριση ανάμεσα στο Sinn Féin και τον, και τον Ήρα. Ε, είναι ελάχιστη η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές οργανώσεις και συχνά χρειάζεται ε, ένα φύλλο σικής, ε, χρειάζεται να προσποιείται κανείς για να έχει διάλογο με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ε, βλέπουμε τώρα το καθεστώ που έχει αποκτήσει τώρα πια το Sinn Féin. Πάντως η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω έχει να κάνει με τις σχέσεις σας με τη Ρωσία. Γνωρίζω ότι το Ισραήλ έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό πληθυσμού ρωσικής καταγωγής. Ο Πρωθυπουργός σας επανειλημμένα έχει συναντήσει τον κύριο Πούτιν. και φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι επαφέ. Μήπω μπορείτε να μα πείτε περισσότερα σχετικά με τη σχέση αυτή. Η Ρωσία μήπω παίζει διπλό παιχνίδι, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στο Ιράν και είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της χώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς βλέπετε εσείς αυτές τις σχέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πασκάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντίχτερ, θα ήθελα καταρχάς ε, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για ε, τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους. Θα πρέπει πάντα να καταδικάζουμε οποιαδήποτε απώλεια ζωής. Ε, πάντως, κύριε Ντίχτερ, πρέπει να πω ότι έχω απογοητευτεί πολύ από την εισαγωγή σας προς την Επιτροπή μας. Γιατί δεν αναφερθήκατε στο κανάλ Αχμετ στην καταστροφή και την παραβίαση του, εθνικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα της ε, τέταρτης ε, σύμβασης ε, της Γενέβης για την καταστροφή της ιδιοκτησίας. Η καταστροφή λοιπόν του Καμαλ Έχμετ μιλώ για τις περιοχές που ελέγχουν οι Ισραηλινοί στην Ιερουσαλήμ και δεν αναφερθήκατε και στη νέα νομοθεσία που δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με ε, τη θέση των Ισραηλινών Αράβων. Γενικά, πώς ε, μπορείτε να αιτιολογήσετε έναν τέτοιο νόμο που ε, θεσπίζει διακρίσεις εις βάρος των Αράβων. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να υπερασπίσετε τη χώρα σας ε, κατά του, της τρομοκρατίας, αλλά θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται ε, συμφιλίωση ε, και διάλογος. Δεν πρέπει πάντα απλά κανείς να προβάλλει τις δικές του θέσεις. Νομίζω ότι οι ανησυχίες των συναδέρφων μου είναι γιατί παραβιάζεται τόσους διεθνείς κανόνες γιατί θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείτε το διεθνέ δίκαιο. Έχετε μια δημοκρατική χώρα στη Μέση Ανατολή, όπου δεν υπάρχουν πολλέ δημοκρατικέ χώρε. Ωστόσο, το δημοκρατικό σα σύστημα δεν φαίνεται και πολύ δημοκρατικό λόγω των ενεργειών τη κυβέρνησή σα και των αρχών σα. Ευχαριστώ, κύριε Καν. Η κυρία Φώτηγα και ο κύριος Οστρεβίσιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Δίχτερ, καλώς ορίσατε την ΑΦΕΤ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με, τον, με τις ανησυχίες του κ. Φανόρντεν για τη Ρωσία, αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για να σας ρωτήσω κάτι για την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν. Η ισχύς, μάλλον συγγνώμη, ε, ποια είναι η θέση σας για τις ε, λαϊκές και στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και τις διαδηλώσεις. Επίσης, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον του Άσαντ στη Συρία μετά τις τελευταίες πρόσφατες ε, εξέλιξεις και ποια ε, είναι η αξιολόγηση σας για την κατάσταση στην Ιντλιμπ. Ο κ. Στραβίσιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Δίχτερ, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε επαφή και να λαμβάνει η χώρα ένα ανοιχτό και ειλικρινής διάλογος ανεξαρτήτως ε, συνθήκων στις οποίες βρισκόμαστε. Καταρχήν τα συλληπιτήριά μου σε όλε τις οικογένειε που έχασαν τους ανθρώπους τους εξαιτία τρομοκρατικών επιθέσεων πρόσφατα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι η θέση σας για την τάση αύξηση του αντισημιτισμού παγκοσμίω. Τι, πόσα θα επηρεάζουν τις συνθήκες ε, διαβίωσης των ε, Ισραηλών εκτός της χώρας, για παράδειγμα. Δεύτερον, σχέσεις σας με την Τουρκία. Έχουν περάσει από πολλές μεταλλαγές, ε, διακυμάνσεις. Πρόσφατα ακούσαμε πολύ αυστηρές δηλώσεις του κ. Ερντοάν τριμερής διάλογος μεταξύ Ερντοάν, Πούτιν και της ηγεσία του Ιράν είναι, αποτελεί ανησυχία για πολλούς στη Δύση. Πώς μπορείτε να περιγράψετε την κατάσταση των σχέσεών σας με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Thank you, colleagues. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι μάλλον. Πολλές ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε και δηλώσεις σας δώσουμε 10 λεπτά για να απαντήσετε όσο πιο πολλές μπορέσετε. Ίσως είναι αδύνατον αυτό, αλλά τέλος πάντων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις μαζί με τα μέλη της Κνεσέτ που με συνοδεύουν από το Ισραήλ. Θα ήθελα να αναφερθώ στις δηλώσεις που έγιναν, που δεν ήταν ερωτήσεις. 47 χρόνια της ζωής μου καταπολεμώ την τρομοκρατία. Έχω δει πολλά είδη τρομοκρατίας. Στο Ισραήλ, την Δυτική Όχθη, την Λορίδα της Γάζας, στο Λίβανο και σε όλο τον κόσμο. Σε στενή σύνδεση με όλες τις χώρες, μεταξύ αυτών και πολλές χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται εδώ. Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει την τρομοκρατία μόνος του. Ούτε το Ισραήλ μπορεί, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπάνια, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και οι αραβικές χώρες. Γιατί η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Η Αλκάιντα δεν είχε σύνορα. Ο Ισλαμικό, το Ισλαμικό κράτος επίσης δεν είχε σύνορα, προσπάθησαν να δημιουργήσουν το Ισλαμικό Χαλιφάτο, ούτε αυτοί γνώριζαν σύνορα. Και είμαι πολύ περήφανο για όλε αυτές τις μάχες που έχω δώσει εναντίον τη τρομοκρατία. Και λυπάμαι για τις περιπτώσεις που εγώ και εμείς χρειάστηκε να επιχειρήσουμε αλλά αποτύχαμε να μπλοκάρουμε τρομοκρατία και το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν άνθρωποι στην Ισραήλ, στο Ισραήλ και σε γειτονικέ χώρε. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ μέσα υπάρχουν πολλοί που έχουν συμμετάσχει σε πολέμους και σε μάχες, σε αντιτρομοκρατικές επιχείρησεις. Δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς λάθη. Αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκοπό να ε, προκαλέσω βλάβη σε αθώους ανθρώπους. Και, και εγώ έχω επιζήσει από τέτοιες συνθήκες και γνωρίζω πολύ καλά τι είναι αυτό. Ε, ο εβραϊκός λαός έχει υποφέρει πάρα πολλά. Και όταν δημιουργήσαμε το κράτος μας, τότε αυτοί που το δημιούργησαν, αποφασίσαμε ότι το κράτος του Ισραήλ θα είναι ένα κράτος, ένα κράτος έθνος για τους Εβραίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να ζήσει στο Ισραήλ. Αλλά η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ ως κράτος έθνους είναι ε, αποκλειστική για τον εβραϊκό λαό. Αυτό το λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν λέει τίποτα εναντίον τα, των ατομικών δικαιωμάτων οποιοδήποτε πολίτη του Ισραήλ. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, οτιδήποτε. Και σας συστήνω να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το θεμελιώδη νόμο μας. Θα εκπλαγείτε. Όταν μίλησα για τους παραλληλισμούς ε, ανάμεσα στι τρομοκρατικέ οργανώσει της Ευρώπης και της μέση Ανατολή, Έχετε δίκιο, δεν υπάρχουν ομοιότητες. Γιατί ακόμα και ο Ήρα και ο ΕΤΑ μέσα σε όλο αυτό το τρομακτικό τρομοκρατικό σύστημα χρησιμοποιούσαν έναν κώδικα προκειμένου να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και θάνατοι αμάχων δεν πέτυχαν πάντοτε, αλλά στα 47 χρόνια πολεμάω τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή. Στην, ε, την τρομοκρατία μέρους των Αραβικών κρατών και των Παλαιστινίων ποτέ δεν είδα ούτε μία περίπτωση ούτε μία περίπτωση που κάποιο να έστειλε ένα κωδικό για να αποφευχθεί ο θάνατος ενός αθώου ατόμου. Τώρα, για το Ιράν. Και ε, ο κ. Μπαλεύ θα μπορούσε ενδεχομένω να πει δύο λόγια παραπάνω. Είναι για το θέμα του Ιράν, το οποίο είναι το κράτος το οποίο πιο πολύ προσπαθεί να κατασκευάσει όπλα μαζικής καταστροφής. Ε, η συμφωνία η οποία είχε επιτευχθεί απλώς αναβάλει για μερικά χρόνια. Θα ήθελα όμω να δώσω στον κύριο Μπελάβ τον, ε, λόγο αν επιτρέπετε. Πρόεδρε, ε, κύριο Μακάλιστα, να σφαρώ, εσεί έχετε τόση εμπειρία να δίνετε το λόγο κι εσεί. Ε, έχετε το λόγο. Εν συντομία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι είμαι μέλος του κόμματος των εργατικών της Ισραηλινής Αντιπολίτευσης. Και φυσικά έχω πολύ μεγάλη κριτική να ασκήσω στην σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση. Ε, επί πολλών θεμάτων όμως συμφωνούμε όλοι. Το να βλέπουμε το Ιράν ως ένα κράτος που προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Μέση Ανατολή δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ο μόνος λόγος για τον οποίο το Ιράν θέλει να απαγιώσει τις στρατιωτικές του ε, ικανότητες στη Συρία. Ουσιαστικά μιλάμε για πυραυλικά συστήματα μεγάλων αποστάσεων και αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα. Δεν, όλο αυτό δεν έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση και ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο μόνος λόγος που το επιθυμούν αυτό είναι για να έχουν στη διάθεσή τους ένα διακόπτη ώστε να επηρεάζουν την ε, περιοχή πολύ εύκολα εφόσον έχουν εγκαταστήσει τέτοια συστήματα στη Συρία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να θέσω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια ερώτηση προς όλους σας. Ένα πράγμα που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι δύο εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι ζουν υπό φρικτές ε, ανθρωπιστικές συνθήκες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που παρότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν, έχει συμφωνήσει να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, δεν καταφέρνετε να το κάνετε. Διότι πιστεύετε ή θέλετε οι επενδύσεις αυτές να περάσουν να, να εγκριθούν από τον Μαχμουντάμπα από τον Παλαιστίνο πρόεδρο, ο οποίος Παλαιστίνο πρόεδρος δεν θέλει να πάρει τα χρήματά σας και να τα επενδύσει στο λαό του στη Γάζα. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο. Και πρέπει να σας φαίνεται παράξενο και σε εσάς πιστεύω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που κανένα σας δεν έκανε αυτή την ερώτηση. Για ποιο λόγο ο Παλαιστίνιος πρόεδρος δεν θέλει να δεχθεί τα χρήματα που το προσφέρετε εσείς ως επένδυση στη Γάζα για να βελτιωθεί η διαβίωση των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντίχτερ. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Γι' αυτό λίγες προτάσεις. Να απαντήσω στην πολύ σημαντική ερώτηση η δική μου επιτροπή πώς μπορεί να είναι αδερφική της δικής σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό το πλαίσιο ε, και ένα από αυτά είναι το αντιτρομοκρατικό σύστημα. Δυστυχώς με αίμα των ανθρώπων μας, των συμπολιτών μας έχουμε πληρώσει ε, τα, τα μαθήματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν νομίζω ότι κάθε χώρα θα πρέπει να πληρώνει έτσι τα μαθήματα αυτά, αλλά έχουμε ε, συγκεντρώσει πολύ πείρα σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι δικοί σας άνθρωποι του χώρου αυτού και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν από μας πώς μπορούν να σώσουν ζωές. Και μερικές φορές η πύρα δεν αγοράζεται στα καταστήματα, αποκτάται από την καταπολέμηση των τρομοκρατών. Και δυστυχώς είχαμε τόσους, ε, τόσους καμικάζι που πολλά χρόνια χρειάστηκαν για να αποκτήσουμε, να διαμορφώσουμε τη σχετική μεθοδολογία, την οποία μπορούμε να σας χαρίσουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δίχτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι από την Κνέσετ, σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε εδώ πέρα για την ανταλλαγή απόψεων και σας ευχόμαστε καλή παραμονή στις Βρυξέλλες και επικοδομητικές συζητήσεις. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην Ιερουσαλήμ. Ευχαριστώ.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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καθυστερήσει. 12 λεπτά καθυστέρηση έχουμε αυτή τη στιγμή. All those guests to leave our committee room. Θα παρακαλούσα τους προσκεκλημένους να εγκαταλείψουν την αίθουσα και να περάσουμε στο σημείο 7. Και θα ήθελα εισαγωγικά να πω το εξή απευθύνομαι σε όλου τους παρόντες συναδέρφους. Προσπαθώ να προεδρεύω στην Επιτροπή αυτή με όσο γίνεται πιο ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο. Πρέπει να πω όμως ότι ε, λυπήθηκα με αυτό που συνέβη στο προηγούμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Κάθε συνάδελφος έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τι απόψει του ελεύθερα στην Επιτροπή μα. Αλλά ακούσαμε αρκετά σκληρή διατύπωση στη συζήτηση με τους Ισραηλινούς προσκεκλημένους μας. Προτείνω να το συζητήσουμε αυτό στην επόμενη συνεδρία του Διαβηρημένου Προεδρείου. Ενδείχνεται κάτι τέτοιο. Πόσο συχνά έχω δίπλα μου προσκεκλημένο με τον οποίο να μην συμμερίζομαι όλες τι απόψει. Και πόσο συχνά, για παράδειγμα, είχαμε από το Ιράν προσκεκλημένου, θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει παρόμοιε παρατηρήσεις. Προσπαθούμε όμως να σεβόμαστε όλους τους προσκεκλημένου μας, άσχετα ε, από το ποιε είναι οι πολιτικέ τους απόψεις τους. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς στο μέλλον θα αντιμετωπίζουμε προσκεκλημένου και από το Ισραήλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να του αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε όλους τους προσκεκλημένου στην Επιτροπή μας. Ε, πρέπει να πω ότι δυσαρεστήθηκα με αυτό που συνέβη. Άννα Γκόμε, ωραία, έκανε τις παρατηρήσεις του, σου, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Απλά θα ήθελα να πω ότι είπατε ότι είναι τιμή σα. Εγώ είπα ότι δεν, δεν ένιωθα τιμημένη με τον συγκεκριμένο προσκεκλημένο και νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό. Ναι, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτά που είπες εσύ, αλλά ε, είπα ότι στο όνομα της ΑΦΕΤ λέω ότι ε, είναι τιμή μας που έχουμε προσκεκλημένους από την ΚΝΕΣΕΤ, όχι μόνο εκείνον. Και αν αρχίσουμε να ε, κάνουμε διακρίσεις, τότε ε, είναι μια μακρά συζήτηση. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τιμούμε όλους τους προσκεκλημένους επιτροπείς Επιτροπής μας. Περνάμε στο σημείο αυτά της ημερησίας διάταξης, έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο και δίνω, ε, για την Αλβανία και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αύριο θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα πρώτα να αναφέρω κάποια θέματα που συζητήσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, σκιώδους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές που σε λιγότερο από μία ώρα ε, καταλήξαμε σε συμβαστικές τροπολογίες και το λέω αυτό διότι είναι καλό δείγμα του ότι επί της αρχής συμφωνούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάποια βασικά μηνύματα. Εδώ και τέσσερα χρόνια η Αλβανία επισήμως έχει αναγνωριστεί ως ε, χώρια υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιστούμε σαφές ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην πραγματικότητα. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τις διαπραγματεύσεις με την Αλβενία. Ταυτόχρονα ε, λαμβάνουμε γνώση της ε, απόφασης του Συμβουλίου του Καλοκαιριού σχετικά με την ε, έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του χρόνου τον Ιούνιο. Λοιπόν, περιμένουμε να ε, ληφθεί η σχετική απόφαση και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Φυσικά, στην, ε, στην έκθεση αυτή, από τη μία, αναφέρουμε τους τομείς όπου είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Από την άλλη, επισημαίνουμε και το τι περιμένουμε από τους ε, Αλβανούς φίλους μας. Το σημαντικότερο σε όλες τις μεταρρυθμίσεις είναι ότι το σημαντικό δεν είναι να ικανοποιήσει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ε, ε, πρόεδρό της, αλλά να βελτιωθούν οι συνθήκες των ανθρώπων στην χώρα. Συμφωνούμε με την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και χαιρόμαστε που βλέπουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Είδαμε πρόοδο στον δικαστικό τομέα και βλέπουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, αυτές αποτελούν και αποτρεπτικό παράγοντα για το μέλλον. Θέλουμε περισσότερη καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, το ίδιο ισχύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, σημαντική πτυχή είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας για τα οποία μιλάμε συνεχώς και θα πρέπει να δούμε εφαρμογή ε, των δεσμεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική τους αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Συμφωνήσαμε να μην αναφέρουμε κάθε μειονότητα, διότι έχουν διαφορετικό μέγεθος, ε, έχουν διαφορετικά προβλήματα, αλλά τα δικαιώματα των μειονοτήτων ισχύουν για όλες. Επίσης, ε, αναφέρουμε την περιβαλλοντική πολιτική και αναφέρουμε ότι όχι μόνο στον ΑΟ ποταμό, αλλά και αλλού θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Και για να κλείσω με κάτι θετικό, Η πολιτική γειτονία αποτελεί σημαντικό θέμα στις συνομιλίες μας με τους Αλβανούς συναδέλφους μας. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλουμε προσπάθειες για σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Οι Αλβανοί το κάνουν αυτό, ευτυχώς δεν το κάνουν μόνοι τους και άλλοι συμμετέχουν στις προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους κοιόδης και περιμένω την ε, ψηφοφορία αύριο και πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης για την Αλβανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κνούτ Φλέκενστάιν για τις εξηγήσεις αυτές. Ε, περνάμε στη συζήτηση. Ο Έντουαρτ Κούκαν από το Έλκιν, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλή συνεργασία προφανώς. Ιδιαίτερα χαίρομαι για τη συνεργασία του κ. με τους κοιόδης ηγητές. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ισορροπημένο και νομίζω ότι θα υπερψηφιστεί χωρίς σημαντικά εμπόδια. Με αυτήν την έκθεση στέλνουμε τέσσερα μηνύματα στην Αλβανία, πιστεύω. Πρώτον, η Αλβανία έχει σημειώσει πρόοδο στη διαδικασία ένταξης και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων του χρόνου. Αυτό ε, θα αναφερθεί και με τροπολογίες. Δεύτερον, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και η δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και να εντοπίσουμε προβληματικούς τομείς. Επίσης να επενέσουμε τις επιτυχίες. Τρίτον, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η αλβανική κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς που σε μεγάλο βαθμό εμποδίζουν την πρόοδο της χώρας. Θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα, όπως επίσης και στο θέμα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, της καλλιέργειας ναρκωτικών και της, ε, του εξοπλήματος ε, χρημάτων. Επίσης, η πόλο στην πολιτική ζωή μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο. Για παράδειγμα, η, ε, οθέτηση των συστάσεων του ΟΑΣΕ από τις τελευταίες εκλογές κόθησε επίσης και ο νέος εκλογικός νόμος αποτελούν σημαντικά βήματα θα πρέπει να καταστεί σαφές στην Αλβανία ότι περιμένουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών. Μία ακόμα φορά ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης της Αλβανίας, αλλά και ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. E ο κ. Τάνοκ για το ECR. Εκ μέρους της ε, κυρίας Θεοχάρου θα ήθελα να διαβάσω αυτή την, ε, την ε, τοποθέτηση. Θεωρούμε ότι τα Βαλκάνια είναι ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία θα πρέπει να συνδεθεί στενά και κάποια στιγμή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά είναι ένα προβληματικό κράτος με σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα κυβέρνηση, τα κόμματα και ο λαός θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορέσουν για να αντιμετωπίσουν την ε, διαφθόρα, να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η έκθεση του κ. Φλέκερστάιν καλύπτει επιτυχώς ε, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την ε, χώρα. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενταξιακή διαδικασία της χώρας. Αλλά δεν θα πρέπει η δημοκρατία να επιβληθεί, θα πρέπει να υιοθετηθεί. Πιστεύουμε ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο και στηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και συνολικά την έκθεση. Ελπίζουμε ότι οι συστάσεις μας θα βοηθήσουν την αλβανική κυβέρνηση και τον αλβανικό λαό να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο να πετύχουν το, την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν από τους Αλβανούς προς συμφέρον τους. Ε, εκτιμούμε όλα τα βήματα που έχουν γίνει ήδη προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζουμε ότι η ελβανική κυβέρνηση θα πρέπει να επιλύσει μέσω του διαλόγου τα προβλήματα που έχει με την Ελλάδα βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις και με σεβασμό των, της ελληνικής και άλλων μειονοτήτων. Κύριε Θεοχάρου, ευχαριστεί τον εισηγητή και την ομάδα του για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Charles Άλντε δεν έχετε ζητήσει να μιλήσετε. Πάμε στους πράσινους εγκοσόλτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον γιατί Είναι εξαιρετική η έκθεση. Πραγματικά η Αλβανία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Δεν πάβει όμως να εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικότερα στο δικαστικό σύστημα, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια διοίκηση. Καθώς επίσης και σε κάποιους τομείς των δημοσίων συμβάσεων. Υπάρχει και το θέμα της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος, θέματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. και που χρήζουν της προσοχής μας για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, εδώ βρισκόμαστε και για να ενθαρρύνουμε τα πολιτικά κόμματα να θεωρήσουν αυτή την ε, διακομματική συνεργασία ως μια ευκαιρία ε, συνεργασίας για να πλησιάσουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή ένταξη ε, μέσω των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την συμπερίληψη της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνίας των πολιτών στις συμβιβαστικές τροπολογίες της έκθεσης. Όπως είπε και ο εισηγητής σε πολλές παλιότερες εκθέσεις, είχαμε αναφέρει αυτό το πρόβλημα του ΑΟΥ και των υδροελεκτρικών εργοστασίων. και οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υποβαθμίζεται εδώ η περιοχή περιβαλλοντικής ε, προστασίας ε, πρέπει να το δούμε βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Πρέπει να ζητηθεί λοιπόν από την αλβανική αρχή να τηρούνται αυτοί οι διεθνείς περιβαλλοντικοί κανόνες. Και τέλος, είμαι βέβαιος ότι η Αλβανία είναι μια χώρα γεμάτη ευκαιρίες πολλές από τις οποίες ε, ε, εναπόκεινται στα χέρια των Αλβανών πολιτικών. Αλλά από την άλλη είμαι βέβαιος ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παράσχει μεγάλη βοήθεια προς την Αλβανία ώστε να σημειώσει πρόοδο και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Ο κύριος Επιτίδιος, παρακαλώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το γεγονός ότι στην έκθεση αναφέρεται η απέτηση προς την αλβανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θετική διότι η μεγαλύτερη μειονότητα που υπάρχει στην Αλβανία είναι η ελληνική μειονότητα της οποίας τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον καταπατώνται. Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνω ότι θεωρώ θετική την ε, τοποθέτηση του εισηγητού να σεβαστεί η αλβανική κυβέρνηση τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ένα σημείο όμως το οποίο δεν συμφωνώ με τον εισηγητή είναι το γεγονός ότι η Αλβανία καταβάλει προσπάθειες για να δημιουργήσει σχέσεις καλής γειτονίας. Είναι γνωστό, έχει αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, το ότι η Αλβανία εγείρει εδαφικές απαιτήσει από όλες τις γειτονικές χώρε τη Ελλάδο μη εξορουμένη. Εάν δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση και αν δεν υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. Κλείνει εδώ λοιπόν η συζήτηση θα ακολουθήσει η ψηφοφορία ως επόμενο βήμα αύριο στις 2.30. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 8, έκθεση της, ε, για την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο και δίνω το λόγο στον κύριο Τσάουτ Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα παραμείνω σύντομος. Ε, Έχουμε τη δεύτερη εξέταση αύριο, όπως σας είπα, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και οδησυγητές ε, για τη θετική του συμβολή. Όπως συνήθως έχουμε επιτύχει ε, καλές συμβαστικές τροπολογίες για τα σημαντικότερα ζητήματα. Αυτό ε, δηλώνεται εδώ και η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί στο Μαυροβούνιο. Λίγα είναι τα διακυβεύματα αναφέρεται στη ελευθερία των μέσων και η καταπολέμηση της διαφθοράς ως βασικές μας ανησυχίες ε, στην έκθεση. Πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλα αυτά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου στον τομέα αυτών. Το επόμενο άλμα θα είναι σημαντικό αλλά δύσκολο, αλλά με βέβαιο ότι το Μαυροβούνιο θα τα καταφέρει. Τώρα απαιτούνται περισσότερα βάσει της ε, διαδικασίας ε, διεύρυνσης ε, και καθώς προχωρά η διαπραγματευτική διαδικασία χρειάζεται να ολοκληρωθούν τα κεφάλαια 23 και 24. Δυστυχώς αυτή θα είναι η τελευταία μου έκθεση ως εισηγητή αυτού του κοινοβουλίου μόνιμου εισηγητή μετά από 10 χρόνια δυστυχώς λόγω του Brexit. Παρότι είμαι σίγουρος ότι το Μαυροβούνιο θα είναι πιθανότατα η πρώτη χώρα που θα αντικαταστήσει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο ως 28, 28ο ε, μέλος μετά από την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα μου δώσει λίγη παρηγοριά σε αυτή την καταστρεπτική πορεία που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η χώρα μου. Τέλο, ε, θα ήθελα να τονίσω τι ε, τροπολογισμού μου 39-40 για την παράγραφο 10 που αντικατοπτρίζουν μια εκ των πραγμάτων αλλαγή ε, και πέραν όλων των συμβασμών, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να τις υποστηρίξουν οι συναδελφοί και θα μου πούν εκ των προτέρων αύριο αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνονται οι παρατηρήσεις μου και σα ευχαριστώ όλου σα για τη συμμετοχή σα σε εκθέσεις αυτές, όχι μόνο σε αυτήν εδώ, σε όλες τις εκθέσεις για το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ Τσάρλ Στάνοκ και εκ μέρους των συναδέλφων ευχαριστούμε για τις καλές σας προσπάθειες ε, ε, και εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τις υποθέσεις του Μαυροβουνίου. Δύο ε, έχουν ζητήσει να μιλήσουν, ο κύριος Αντέμοφ, ο κύριος Κούκαν και ο κύριος Ράντος του κύριο Σόλτες, Φλέκενστάιν. Ωραία λοιπόν. Ξεκινάμε με τον κύριο Αντέμοφ εκ μέλους ε, ε, του κύριου Αντρέη Κονάτσεφ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να μεταφέρω τη συγγνώμη του κύριου Κόβετσεκ ε, για την απουσία τη βρίσκεται στο Ισραήλ ως αντιπρόεδρος, αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΕΛΚ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσει τον ε, κύριο Τάνοκ για την επικοδομητική δουλειά που έχει κάνει πάνω στην έκθεση αυτή. Στην έκθεση αυτή και στις και στις σχετικές ε, τροπολογίες είναι απόλυτα συνεπείς. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή αναγνωρίζουν τα βασικά προβλήματα. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ε, της καταπολέμησης της νομοποίησης ε, παράνομων εσόδων, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το καθεστώς της δημόσιας τηλεόρασης και η κατάσταση των δημοσιογράφων. Οι συναντήσεις με τους κοιόδες εισηγητής ήταν πολύ επικοδομητικές και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι το τελικό κείμενο είναι πολύ ισορροπημένο και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν. Νομίζω ότι το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει ε, ιδιαίτερη πρόοδο και καλό όλους να το αναγνωρίσουν αυτό. Υπάρχουν όμως ακόμη μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέμοφ. Ο κύριος Κνουτ Φλέκενστάιν πολύ σύντομη. Ο κύριος Ανδρουλάκης και ο συζητητής μας δεν μπορεί να είναι παρόν και απλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε ευγνώμονες για την πολλή δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Τάνοξ. Συμφωνούμε μαζί του και τον ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία του με τους κοιόδης συζητητές. Θα υπερψηφίσουμε αύριο την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κνούτ Φλέκενστάιν. Ο κύριος Ράντος από την Άλτε. Δεν είστε στο Σαραγεύο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ όχι μόνο για την καλή συνεργασία στην έκθεση αυτή, αλλά και στην δουλειά, τη συνεργασία μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και για την δική του δουλειά τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την αισιοδοξία του την οποία πάντα εκφράζει όταν μιλάμε για την προσχώρηση του Μαυροβινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αρκετά σταθερή η πρόοδος, αν και αργή. Υπάρχουν δυσκολίες σε βασικούς τομείς οι μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί πολύ αργά ε, στον τομέα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της ε, καταπολέμησης ε, της διαφθοράς, της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ωστόσο, η μόνη προοπτική για το Μαυροβούνιο και τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι η προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει πολύ θετικά μηνύματα με την έκθεση αυτή. Αυτή την οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόλτες από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή συμβαστική πρόταση και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ε, για την ε, παράγραφο 28, τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, στην παράγραφο 28 έχουμε πολύ σαφή διατύπωση σχετικά με το πρόβλημα ε, της Ουλσίν Σαλίνα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω στο θέμα των ε, επενδύσεων ε, και έχουμε και την τροπολογία μας ε, σχετικά με την λίμνη ισκαγκα Όσον αφορά την διαφθορά, θα ήθελα επίσης να συστήσω συναδέλφους να υπερψηφίσουν την τροπολογία 25, καθώς και την τροπολογία 69 σχετικά με τον Οργανισμό Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Ξέρουμε ότι ε, είναι πολύ επώδυνα τα μέτρα αυτά για κάποιους στη χώρα. Ε, αναπτύσσεται όμως μια πολύ καλή ε, και ζωντανή δημοκρατία στο Μαυροβούνιο και δεν θα πρέπει να τεθούν εμπόδια στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες. Η ΓΚΟΕ, η FTD, η ΕΝΕΦ, κανείς δεν είναι παρόν. Έντουαρτ Κούκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος, διότι συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο κύριος Κόβατσεφ, ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Εκτιμώ τη δουλειά του Τσάρλ Στάνοκ και τον ευχαριστώ για την πολύ ε, επαγγελματική και ικανή δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Το Μαυροβούνιο προοδεύει σταθερά με την υποστήριξη των πολιτών. Απομένουν κάποια πράγματα να γίνουν στην διαδικασία της μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και την επιβολή του κράτους δικαίου. Ε, χρειάζεται να καταδικάσουμε απερίφραστα ε, τα φαινόμενα εκφοβισμού, ε, συκοφαντίας δημοσιογράφων. Καλούμε τις αρχές να εξετάσουν τις ε, σχετικές υποθέσεις. Επίσης είναι ε, κρίσιμη σημασία η ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Επίσης είδαμε το ε, μποϊκοτάρισμα στο Κοινοβούλιο του Μαυροβινίου, αλλά θα ήθελα να επενέσω το Μαυροβούνιο για την ευθυγράμμιση με την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Το Μαυροβούνιο βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση από κάποια τρίτη χώρα, γι' αυτό θα πρέπει να επενέσουμε ακόμη παραπάνω τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Κούκαν, ο Τσάλ Στάνοκ για να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν ένα από τα πιο ωραία αποχαιρετιστήρια δώρα από τους συναδέλφους μου εδώ πέρα σύντομα και ε, καλά. Ε, Σα ευχαριστώ για την εκτίμηση τη δουλειά που έχω κάνει. Σημειώνω τι παρατηρήσει του Έντουαρτ Κούκαν σχετικά με τον εκφοβισμό δημοσιογράφων και την ε, ελευθερία του τύπου. Νομίζω ότι αυτά καλύπτονται επαρκώ στην έκθεση. Επίση, συμφωνώ με του πράσινου όσον αφορά τι περιβαλλοντικέ ανησυχίε σε προηγούμενε εκθέσει. Κατά τα άλλα, είναι ε, μία από τις λίγες εκθέσεις που στηρίζονται από, πολλά πολιτικά, από πολλές πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και ελπίζω ε, το Μαυροβούνιο τα επόμενα χρόνια να προσεγγίσει όλο και περισσότερο την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ, Charles Τάνοκ. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης. Θα ψηφίσουμε αύριο το μεσημέρι εδώ στην ΑΦΕΤ. Και φτάνουμε στο επόμενο θέμα, το υπαριθμό 9. Εξέταση των τροπολογιών ε, τη έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπή του 2018 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δίνω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Βάγγλ, που θα μας παρουσιάσει τα επόμενα βήματα. Παρακαλώ, Ήβο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι θα μιλήσω στα σλοβενικά. Οπότε, αν θέλετε, βάλτε τα ακουστικά σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες τις συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι πιο ενθαρρυντική, πιο ανοιχτή, πιο θετική από ό,τι τα προ... τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τους Έλληνες συναδέλφους για αυτή την επιτυχία. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις των Σκοπίων και των Αθηνών ενέπνευσε πολλή αισιοδοξία σε όλους εμάς. Περιμέναμε για πολύ καιρό και ελπίζουμε ότι αυτή η περίοδος αναμονής θα τελειώσει. Αναμένουμε τα Σκόπια να ξεκινήσουν τη διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της ε, διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η, Μακεδονία, λέει ο Μιλτής, προσπαθούσε να ξεφύγει από την πολιτική κρίση που τη μάστιζε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. ε, συνεισφέραμε και στο διάλογο Ζαν Μονέ και στη Συμφωνία Πρεσνό. Ο διάλογος Ζαν Μονέ μάλιστα ακόμα συνεχίζεται. Μετά την υιοθέτηση αυτής της έκθεσης και αφού η Μακεδονία επιλύσει τη νέα πολιτική κρίση που δημιούργησε το δημοψήφισμα κατά, τη διάρκεια, ε, κατά την άποψη κάποιων ήταν επιτυχημένο, κατά την άποψη κάποιων άλλων όχι. Μετά από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, για αφού λυθεί αυτή η πολιτική κρίση, θα υπάρχει και πάλι πολύ έργο μπροστά μας. Θα πρέπει οι ίδιοι να υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτημένο σε όλους τους τομείς. Και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το εξής. Θέλω να ζητήσω από όλους να στηρίξουν την προφορική τροπολογία που έχω υποβάλει. Περιμένουμε να γίνουν πρόσθετα βήματα εκ μέρους της κυβέρνησης Μακεδονίας και είτε με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο είτε με την την προσφυγή σε εκλογές προκειμένου να, αν δεν, μπορέσει να επιτευχθεί λύση με το παρόν κοινοβούλιο. Το σημαντικό όμως είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Μακεδονίας να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ υπό την προπιβόθεση ότι αυτή είναι η επιθυμία της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι, όπως και οι άλλες χώρες και για τις άλλες χώρες έχουμε Είπατε Πέτερλε, είναι ο κύριος Βίβο Βάγκλο, ο συνάδελφος που είναι συγητής, ε, έκανε λάθος ο πρόεδρος. Θέλω να μιλήσουν Κούκαν, Φλέκενστάιν, Τάνοκ, ε, κυρία Σακοράφα, κύριος Επιτίδιος, και Κούλογλου. Φυσικά σας γνωρίζω, λέει ο Πρόεδρος. Άλλοι Έλληνες συνάδελφοι. Ξεκινάμε τον Έντουαρτ Κούκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ο κύριος Βάγκελ έδειξε μεγάλη ευθύνη ως εισηγητής. Η έκθεση του είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς ε, μελέτης του κειμένου, εξέτασης των τροπολογιών συνεργασίας με τους κοιόδης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Σε σχέση με το θέμα αυτό, την περασμένη εβδομάδα ήμουν στη Σόφια, όπου έγινε μια συνάντηση κοινοβουλίων από όλε τι ε, χώρες ε, των Βαλκανίων και η κατάσταση στη χώρα που συζητήθηκε είναι δραματική. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ιβο για τι περαιτέρω εξέλιξει μετά από το δημοψήφισμα. Την εξολογούμε. Το μόνο που έχω να παρατηρήσω εγώ είναι ότι εάν χρειαστεί να γίνουν πρόορες εκλογές, η χώρα θα οδηγηθεί σε χάος για πολύ καιρό. Συμφωνώ λοιπόν με την τροπολογία που υποστηρίζει να πάμε να ψηφίσουμε αύριο το ψήφισμα. Προλαβαίνουμε πριν από την Ολομέλεια για επικαιροποίηση ανάλογα με τις εξελίξεις στη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Έντουαρτ Κούκαν. Κνούτ Φλέκενστεν, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. κύριε Βάγγελ, συνάδελφοι, αγαπητοί Συνάδελφοι, μιλώ εδώ εκ μέρου του κυρίου Πέτερλε. Είχε κάποιε δυσκολίε με την πτήση του. Θα έρθει αργά το βράδυ. Εκ μέρου του, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και για την καλή συνεργασία. Υποστηρίζω την απόφαση του να ψηφίσουμε αύριο. Ξέρω ότι κάναμε μια συζήτηση για το ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο, αλλά συμφωνώ, ειδικότερα με την προφορική τροπολογία, ότι ακριβώ αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ δυστυχώς λυπάμαι για το αποτέλεσμα. του δημοψηφίσματος δεν ήταν ό,τι είχαμε επιθυμήσει σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση βασίζεται σε πιστικά αποτελέσματα και στην υποστήριξη της αντιπολίτευσης με τόσο μικρή προσέλευση. Ελπίζω η συμφωνία για το όνομα να μην είναι ένα παράπλευρο θύμα τη ευρύτερη πολιτική κρίσης που ανοίγει και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών όπως είπε ο κύριος Κούκαν ήδη. Τώρα, όσον αφορά την εκθέση πρόοδου, που ψηφίζουμε αύριο, στην περίπτωση της Μακεδονίας πέρυσι, μπορούμε να μιλήσουμε για πρόοδο. Έχει την καλύτερη πρόοδο από όλες τις χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρέχουσα κυβέρνηση δεν είχε ένα εύκολο έργο μετά από πολλά χρόνια απουσίας πρόοδου, μάλλον το αντίθετο από την πρόοδο. Η έκθεση επενεί τις προόδους και την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη γείτονα χώρα, με τις γείτονες χώρες, με τη Βουλγαρία και με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι το πολιτικό κλίμα στη χώρα γενικότερα ανοίγει περαιτέρω επικοινωνία με τους πολίτες και υποστηρίζουμε αυτή ε, τη φιλοσοφία διαλόγου αυτό φυσικά δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αποδίδεται στην κυβέρνηση, αποδίδεται και στον νέο αρχηγό της αντιπολίτευσης και στο δικό του κόμμα. Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε τι απομένει ακόμα να γίνει. Να ξεκινήσουν επιτέλους ε, κάποιες σημαντικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του πολιτικού κλίματος στη χώρα γενικότερα με πιο ανοιχτή επικοινωνία και υποστήριξη ε, του διαλόγου. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ε, μεταρρυθμίσεις περαιτέρω, μεταρρυθμίσεις ε, στον οικονομικό, το δικαστικό τομέα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να γίνουν πιο ελεύθερα και για να καταπολεμηθεί επίσης η διαφθορά. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει το πολιτικό της θάρρος ε, για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, μετά από το δημοψήφισμα, πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε πλήρη υποστήριξη. Ελπίζουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις του χρόνου. Ευχαριστούμε ξανά για τη συνεργασία του τον εισηγητή. Πιστεύω ότι το κείμενο είναι ικανοποιητικό και ε, πιστεύω ότι η αυριανή μας ψηφοφορία θα δείξει ευρεία υποστήριξη προς την έκθεση και στο λαό της Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Thank you, Knut Ευχαριστούμε Knut Fleckenstein για το ECR ο Charles Θάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους ε, ε, είναι πολύ καλή η έκθεση του Ιβο Βάγκλ και ελπίζω ότι θα εγκριθεί μετά από τις διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ωστόσο, η συμβαστική τροπολογία 5 που σχετίζεται με το δύσκολο ζήτημα του ονόματος είναι κλειδί για την πρόοδο. Χωρίς επίλυση αυτού του προβλήματος η διαδικασία προσχώρησης της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στα χαρτιά μετά από το δημοψήφισμα στι 30 του προηγούμενου μήνα είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Ωστόσο οι εξελίξει ε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν ότι δυστυχώς η συμφωνία μπορεί να μην υλοποιηθεί λόγω της χαμηλής προσέλευσης που δεν έφερε το 50%. Και τώρα έχουν ξεκινήσει και ομιλίε και φήμε για νέε εκλογέ. Όπω είπε ο εισηγητή του ΗΠΑ, ο Μαθηνή ότι μπορεί να χρειαστούν άλλα 25 χρόνια μέχρι να έχουμε μια νέα συμφωνία, αν χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία. Αυτό θα ήταν τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά για ολόκληρη την ατζέντα τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, το ΕΣΕΑΡ υποστηρίζει το γενικό ο πνεύμα τη έκθεση και τη προσπάθεια τη νέα κυβέρνηση και ειδικότερα το γεγονό ότι εστιάζεται στην ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση ε, στο κράτο δικαίου, των ελευθεριών, των μέσων μαζική ενημέρωση, στην καταπολέμηση τη διαφθορά, αλλά και για την ανάπτυξη ε, καλύτερων σχέσεων στη γειτονία με τη Βουλγαρία, ειδικότερα και την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Ιβο Βάγγελ για τη θετική του προσέγγιση ως εισηγητή και για τις προσπάθειες του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Thank Charles. Ευχαριστώ, Τσάρλς. Ίγκο Σόλτες. Ε, Συγγνώμη για την ΚΟΕ, η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγκλ για τη δουλειά του και επίσης ε, να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο κείμενο. Όμως η συμβαστική που αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών με βρίσκει αντίθετη για λόγους ουσίας κύριε Πρόεδρε. Αυτό το νομικό τεχνοκρατικό δημιούργημα είναι πολιτικά αναφάρμοστο. Πρόκειται για τεχνικό κατασκεύασμα κατά παραγγελία εξωγενών παραγόντων που αδιαφορεί αν διαωνίζεται χρόνια προβλήματα των δύο χωρών αλλά αδιαφορεί και για τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά στη διαδικασία, ο τρόπο και ο βαθμό τη ομής παρέμβαση από όλου σχεδόν του αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακυρώνει στην πράξη τη μεγαλοστομίας τη Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοκρατία και σεβασμό στη θέληση των πολιτών. Και αυτό το τιμωρούν οι πολίτε, ανεξάρτητα αν αρέσει ή όχι. Συνέβη στο δημοψήφισμα τη Ελλάδα, επαναλήφθηκε στο Brexit και με μεγαλύτερη ένταση τώρα στην Φύρον με τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέπουμε του πολίτε να αντιδρούν, να γυρίζουν την πλάτη και να απαξιώνουν όλε τι σοφέ νοθεσίε. Και πάλι, παρόλα αυτά, βλέπουμε του αρμόδιου να συνεχίζουν να πιέζουν, δείχνοντα περιφρόνηση για τη στάση των πολιτών. Με τέτοιε πολιτικέ συμπεριφορέ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να απορούμε για την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών αλλά και τη άκρα δεξιά. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η δημοκρατία σημαίνει πειθό μέσω του διαλόγου και σεβασμό στην πλειοψηφία. Όχι μονόλογο, όχι απειλέ, αλλά και περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών. Η τακτική ακολουθείται σήμερα και στην Ιταλία, από ό,τι βλέπουμε. Η μονομερή αυτή τακτική, κύριοι συνάδελφοι, το έχω ξαναμπεί πάρα πολλέ φορέ, μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει για το μέλλον τη Ευρώπη. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τι συμπεριφορέ μα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Thank you. Would you accept the blue... Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε την ε, γαλάζια κάρτα του κυρίου Φλέκενστάιν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Ότι ο κύριος Φλαγκεστάιν είναι ε, απέναντι και αντίθετο με την Ελλάδα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, την προηγούμενη φορά μα είχε προσβάλει βαθύτατα μέσα στην Επιτροπή. Ότι εμεί οι Έλληνε έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά την πατρίδα μα, την πατρίδα μας, τη χώρα μα και προσπαθούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά τη. Με τον τρόπο που εμεί πιστεύουμε. Ο κ. Φραγκεστάιν πιστεύει άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να δω την ερώτησή του. actually uh, giving Mr. Fleckenstein the blue card was supposed to be a slightly humorous. Ε, ναι, ε, αστειευόμουν όταν ε, ρώτησα αν δέχεσαι την γαλάζια κάρτα, αλλά μάλλον δεν είναι η κατάλληλη μέρα για χιούμορ στην Επιτροπή μας. Κνούτ, επιμένεις να σχολιάσεις. Θα αφήσω το όνομά σου στον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε δύο ακόμη ομιλητέ και μετά θα δώσω το λόγο. Κύριο Επιτίδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δημοψήφισμα το οποίο έγινε στα Σκόπια την προηγουμένη εβδομάδα είναι άκυρο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 73 του συντάγματος τη χώρα, δεν συμμετείχε σε αυτό το 50% των ε, εχόντων τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Κατά συνέπεια, ό,τι έγινε είναι ως μη γενόμενο. Πέραν αυτού όμως, το γεγονό και μόνο ότι πραγματοποιήθηκε αυτό το δημοψήφισμα ικανοποιεί και δικαιώνει τι θέσει των Ελλήνων πατριωτών ότι η διαμάχη της Ελλάδος με τα Σκόπια για το όνομα ήταν εκείνη η οποία ευθύνεται για την μη ευόδοση των προσπαθειών της χώρας αυτή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κατέρευσε πλέον αυτό το άλοθη, όλοι αντιλαμβάνονται ότι η περαιτέρω πορεία των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά θέμα δικής τους αρμοδιότητας και δικής τους ευθύνης. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Thank you, President. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ χρήσιμο και θετικό το ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την συμφωνία που δίνει τέλος σε αυτή την γελία διαφορά για το όνομα και δεύτερον φέρνει σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων περιοχή η οποία μαστίζει τα πολλά προβλήματα. Χτες, δίπλα στα Σκόπια, στη Σόφια, και σε μια άλλη πόλη μάλλον της Βουλγαρίας δολοφονήθηκε μια Βουλγάρα δημοσιογράφος. Επίσης έχουμε την ε, διαφορά ανάμεσα στους Σέρβους και τους Κωσοβάρους για μια τεχνητή λίμνη κλπ. κλπ. Χρειάστηκε πολιτικό θάρρος και από τις δύο πλευρές. για να συναυθεί αυτή η συμφωνία. Γιατί και στις δύο χώρες υφίσταται μια δημαγωγική, εθνικιστική αντιπολίτευση σε αυτή τη συμφωνία. Με μια συμμαχία μεταξύ των φασιστών και της δεξιάς κυρίως. Στην Ελλάδα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται σε αυτήν την αντιπολίτευση. Περιμέναμε μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση της δεξιάς. Από τους εθνικιστές ή από τους νεοναζί όχι ενδεχομένως, αλλά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ναι. Θα ήθελα τέλος να πω ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Ζάεφ αξίζουν μια διεθνή αναγνώριση για το πολιτικό θάρρος που επέδειξαν να συνάψουν αυτή τη συμφωνία που δίνει τέλος σε μια μακρόχρονη διένεξη. η οποία είχε τους ιστορικούς της της λόγους προφανώς, αλλά φορούσε και ένα όνομα. Κύριε Φλεκενστάιν, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Hey, Ευχαριστούμε. Θα ήθελα κάποιο άλλο να μιλήσει. Κύριε Φλέκενστάιν, παρακαλώ, μπορείτε να μιλήσετε. Ich wollte nur zwei Dinge sagen. Δύο πράγματα ήθελα να πω. Καταρχάς, αν έχω προσβάλει κανέναν ή αν έχω προσβάλει την Ελλάδα, ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου και ευχαρίστω να συζητήσουμε πώ θα μπορούσα να εκφραστώ διαφορετικά, να το διατυπώσω διαφορετικά. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, διότι η συμφωνία θα. Ε, θα ε, υποβληθεί στο ε, Κοινοβούλιο και γι' αυτό είναι μάλλον θεωρητικό το ερώτημα ε, αν ήταν επιτυχές ή όχι το αποτέλεσμα. Και τέλος, δεν ξέρω αν ήταν η δική σας άποψη ή αν ήταν η άποψη των πρασίνων. Πολύ θα με ενδιαφέρει να ξέρω πώς θα ψηφίσουν οι πράσινοι αύριο, διότι μιλάμε για την έκθεση και δεν μιλάμε για το δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε πώς θα ψηφίσετε αύριο. Οι πράσινοι μπορούν να απαντήσουν πώ θα ψηφίσουν αύριο πάνω στην έκθεση αυτή. Δεν έχουμε πράσινο στην αίθουσα. Υπάρχει κάποιο σύμβουλο των πρασίνων που θα μπορούσε να μιλήσει με τον κύριο Φλέκενστάιν. Όχι, κανένα πράσινο. Ωραία. Ξαναδίνουμε το λόγο στον Ιβο Βάιγκελ για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλά θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο που επένεσε το θάρρος και τη δημιουργικότητα ε, και των δύο πρωθυπουργών ε, της Μακεδονίας και της Ελλάδας που απέδειξαν ότι με καλή θέληση μπορεί κανείς να ξεπεράσει ιστορικές προκαταλήψεις και να οδηγήσει το χρόνο προς σταθερότητα και αλληλοκατανόηση στα Βαλκάνια. Επίσης θα ήθελα να κάνω κάτι που δεν έκανα πριν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσους επένεσαν το ρόλο του κυρίου Τάνοκ εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Ήτανε μεγάλη χαρά, Charles, να σε ακούμε, διότι πάντα ήταν επικοδομητικά και πολύ καλά προετοιμασμένα τα επιχειρήματά σου. Θα ευχόμουν να παραμείνεις εδώ μαζί μας. Ελπίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτή η πιθανότητα. Ευχαριστώ πολύ και για την καλή συνεργασία. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έτσι, κλείνουμε το θέμα αυτό. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 2.30 η ψηφοφορία. Και περνάμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης και έχω την τιμή να παρακαλέσω τον κύριο Πάσκο να προεδρεύσει στο τελευταίο θέμα της σημερινής ε, ημερησίας διάταξης. Ε, α, όχι, κύριε Κούκαν, Έντουαρτ, παρακαλώ εσύ να προεδρεύσεις. Ε, τουλάχιστον κάποιος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει. Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης, εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Είναι η δεύτερη εξέταση της έκθεσης πάνω στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία και Χωρίς πολλά πολλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ, τον εισηγητή μας, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και να σχολιάσει τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Μίχαηλ, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Ε, το Νοέμβριο θα ψηφίσουμε εδώ στην ε, Επιτροπή μας την ε, έκθεση αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διάφορες σημαντικές συναντήσεις με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης έχουμε το μνημόνιο με τις προϋποθέσεις για το τέταρτο πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας. Θα ήθελα λοιπόν σύντομα να μιλήσω για μια διάσκεψη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, την ε, ε, διάσκεψη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στη Γιάλτα και επίσης έχουμε την ε, συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σολίψης και κατόπιν έχουμε στη Μαριόπολ συνάντηση, είχαμε διάφορες επαφές και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε μια συνάντηση όπου συμμετείχε και η Άννα Είχαμε μια πρώτη συνάντηση κοινοβουλευτικής, ε, της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης με την Μολδαβία και την Ουκρανία. Με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις χαίρομαι που συνεχίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να έχουμε μια σχετικά ευρία συνένεση όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ουκρανίας. Αυτό προκύπτει και από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και από τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν διατυπωθεί. Γενικά, έχω την εντύπωση ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να μην προχωράνε με την ταχύτητα που θέλουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η ε, Ουκρανία προοδεύει και είναι ανοιχτή απέναντι σε αυτά που περιμένουμε εμείς από αυτήν. Υπάρχει το θέμα της παράτασης του ειδικού καθεστώτος σε κάποιων περιοχών ε, στον Τόμπας. Υπάρχουν κάποια, κάποιες κατεχόμενες περιοχές. Πρόκειται όμως για θετική, για θετική εξέλιξη και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε. Παρατηρούμε ότι η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων, για παράδειγμα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συνεχίζεται όπως και άλλες μεταρρυθμίσεις, παρότι είναι αισθητό ο προεκλογικός αγώνας ήδη τώρα. Τον Μάρτιο προβλέπονται προεδρικές εκλογές. Στις ε, συναντήσεις της ε, διακοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης συζητήθηκαν πολλά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας. λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις με τη Ρωσία, όπου δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Από ρωσικής πλευράς, δεν φαίνεται να υπάρχει βούληση για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στις περιοχές που συνορεύουν με τα κατεχόμενα. Η κατάσταση είναι άσχημη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της στα ανατολικά της χώρας. Εκεί προσπαθεί να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων. Όσα, όσον αφορά τις κατεχόμενες περιοχές, δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές αυτές, οπότε δεν μπορεί να αξιολογήσει πλήρως την κατάσταση. οι βουλευτές επιθυμούν και αναφέρομαι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Τυφλίδα. Η επιθυμία των βουλευτών λοιπόν των τριών αυτών χωρών, της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας. Επιθυμία λοιπόν των βουλευτών αυτών είναι να προωθήσουν την εφαρμογή των ε, συμφωνιών. Επίσης έχουμε το νέο ε, πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής των Πρόσκης ε, έχει υπογράψει την σχετική συμφωνία. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι έμαθα για μια μελέτη του συναδέλφου Σόλτς, που λέει ότι η Ουκρανία με πιο αποτελεσματική φορολογική πολιτική θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερους πόρους από τους πλούσιους πολίτες της και ο στόχος αυτός, ε, εάν μπορούσε να επιτευχθεί, θα ε, σήμαινε έσοδα αντίστοιχα με την βοήθεια που παρέχουμε εμείς. Ε, επίσης βλέπουμε ε, διοικητική απλούστευση, 700 συγχωνεύσεις δήμος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αναμένονται και άλλες. Ε, δεν έχουν πραγματοποιηθεί όμως οι δημοτικές εκλογές. Στην ε, συγκεκριμένη περιοχή μένουν ένα εκατομμύριο ε, πολίτες ε, και δεν μπορώ να δεχτώ προεκλογικές υποσχέσει να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα της περιοχής. Ε, έχουν ήδη οριστεί οι αξιωματούχοι όλοι εκτός από έναν και Περιμένουμε να δούμε την πραγματοποίηση των ε, εκλογών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την προσπάθεια αποκέντρωσης με 102 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας είπα, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συζητήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων. Γενικά υπάρχει συμφωνία, η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. και τα οποία δεν θα πρέπει να κολλήσουν λόγω της προεκλογικής διάθεσης. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις που να μπορέσουν να βρουν την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερων συνάδελφων. Το Σαββατοκύριακο λάβαμε μια είδηση από ε, Σιβηρική φυλακή, ο Όλεκ ε, σταμάτησε την απεργία πείνας του μετά από 145 ημέρες. Θα πρέπει να ζήσει για την Ουκρανία και όχι να πεθάνει λόγω του κυρίου Πούτιν. Και εδώ θα ήθελα να κλείσω την εισαγωγή μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. for the very comprehensive introduction. Δίνουμε το λόγο τώρα στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν ο λόγος στον κύριο Πάσκο. Ε, εκ μέρου του ξενόμα του Πίτσουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα παρουσιάσω τη θέση του κ. Πίτσουλα. Καταρχήν θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Γκάλερ και τους σκιώδης Είναι επεπισμένος ότι έχουμε ένα καλύτερο κείμενο πια οι τροπολογίες του αφορούσαν τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης στη χώρα και το να τονίσουμε ότι χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Καταπολέμηση της διαφθοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να παραμείνει ως προτεραιότητα. και η λειτουργία του Εθνικού Γραφείου κατά της διαφθοράς ε, θα πρέπει να στηριχθεί με επαρκείς πόρους. Επίσης, ο κ. Σπίτσουλα τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα των κρατικών φορέων, που είναι κλειδί για την εφαρμογή της συνθήκης, της συμφωνίας μάλλον, αναφέρει την διαβούλευση και έλεγχο της υλοποίησης των, της νομοθεσίας. Ευχαριστεί τελικά τον κύριο Γκάλερ, ο οποίο υιοθέτησε τις περισσότερε από τις εισηγήσει του κύριου Πίτσουλα και ελπίζει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία μέχρι την ψήφιση τη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κ. Τσάλ Τάνο και θεσιά. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκάλερ, πεπειραμένο συνάδελφο. Ο Μακλή και εγώ παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Ουσιαστικά το 2002 ήμουν ένα από του πρώτου που έγραψε στη Wall Street Journal σύσταση ε, ευρωατλαντικής προοπτικής ε, για την Ουκρανία. Τότε ε, έγιναν μάχες στο ΕΛΚ, θα το θυμάστε, που τόλμησα να προτείνω κάτι τέτοιο. Χαίρομαι και λυπάμαι όμως ταυτόχρονα σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα, καθώς έχουν περάσει 15 ή παραπάνω χρόνια. Ουδέποτε τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στην Ουκρανία έστω και πιθανότητα κράτους υποψήφιου και είχε και την πιθανή επιθετική κίνηση από τη Ρωσία με την προσάρτηση της Κρεμαίας ε, με παραβίαση διεθνών συμφωνιών. Τώρα έχουμε μια καλή ε, συμφωνία ε, σύνδεσης ε, και εμπορίου. Η οικονομία υποφελείται από αυτό και από τις παραχωρήσεις τις εμπορικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τέτοιες εποχές πλησιάζοντας το Brexit πολλοί θα έλεγαν ότι θα ήθελαν ενδεχομένως να είχαν μια συμφωνία τύπου Ουκρανίας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θέλω να πω ότι τέτοια συμφωνία δίνουμε στην Ουκρανία για να έρθει πλησιέστερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ε, να πάρει διαζύγιο όπως έκανε η δική μου χώρα. Συγχαρητήρια λοιπόν Μάικλ. Υποστηρίζουμε και εμείς ε, στεναρά την έκθεση αυτή και αναμένω να δω τις ε, τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Very much. I don't see any representatives Δεν βλέπω εκπροσώπηση από τις άλλες πολιτικές ομάδες, οπότε δίνω το λόγο ατομικά σε βουλευτές. Κύριε Μπότσκο, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Καταρχήν, επί του ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν έχει σημειωθεί πρόοδο. Όμως υπάρχουν πολλά ανεπίλητα θέματα ακόμα. Και δεν αναφέραμε ακόμα την προστασία των μειονοτήτων, το οποίο έχω θίξει και έχω συμπεριλάβει σε τροπολογίες εκ μέρους της ε, Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ουγγαρίας. Είναι πολύ σημαντικό να μην μιλάμε μόνο για την για αυτά τα θέματα όταν γίνεται συζήτηση για τη Σερβία του Κωσυφοπέδιου, αλλά και για, όταν μιλάμε για την Ουκρανία. Μειονότητες δεν υπάρχουν μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια. Το θέμα των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εντάσεις που υφίστανται. Προκειμένου η Ουκρανία να προχωρήσει το δρόμο του σεβασμού των διεθνών της υποχρεώσεων. Για μία ακόμα φορά θέλω να αναφέρω το παράδειγμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στις 4 Οκτωβρίου σε πρώτη ανάγνωση υιοθετήθηκε ο νέος γλωσσικός νόμος, όπως ονομάστηκε, που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ουκρανική γλώσσα. Αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει μια εθνική γλωσσική διένεξη. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο στόχος της Ουκρανίας με αυτό τον νόμο, επιβάλλοντας τα Ουκρανικά σε μια χώρα στην οποία υφίστανται και συμβιώνουν διάφορες γλωσσικές μειονότητες. Είναι πολύ σοβαρό. Άλλο ζήτημα, το οποίο εφήγη όμως προηγουμένως, είναι ότι στην Ουκρανία δρούν ακροδεξιές οργανώσεις με αιτήματα όπως για παράδειγμα εκδίωξη της ουγγρικής μειονότητας από την Ουκρανία. Πρόκειται για εξτρεμιστικά αιτήματα τα οποία είναι προφανώς απαράδεκτα. Άλλες οργανώσεις και άλλα μέσα στοχοποιούν συγκεκριμένα άτομα και ζητούν την εξουδετερώσή τους. Η Ουκρανία θα πρέπει να τηρήσει τις, εθνικές της, τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις και γι' αυτό το λόγο και εμείς θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε από κοντά, να βεβαιωθούμε ότι πράγματι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και γίνονται όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βοτσκόρ. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον Μάικλ Γκάλερ και να τον συγχαρώ. Εξαιρετική δουλειά. Ε, όσον αφορά την Ουκρανία, και τη σχέση μας με την Ουκρανία ώστε να μπορέσει η χώρα αυτή να αντιμετωπίσει καλύτερα τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις ειδικότερα όσον αφορά την επιθετική κίνηση της Ρωσίας. Απλά θα ήθελα να προσθέσω και θέλω να τονίσω πόσο ενδιαφέρον είχε η διακοινοβουλευτική συνέλευση στην οποία περιβρεθήκαμε την περασμένη εβδομάδα με αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στη Τυφλίδα και πιστεύω ότι αυτή η διακοινοβουλευτική διάσκεψη μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη και για τις τρεις χώρες, αλλά και για εμάς. Θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε πώς μπορούμε να παράσχουμε καλύτερη βοήθεια για κάλυψη των αναγκών. Δεδομένων αυτών θα ήθελα να υπογραμμίσω έναν τομέα όπου έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει και θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Αναφέρομαι στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά αναφέρομαι στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών στην Ουκρανία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις μας, που ήδη γνωρίζω είναι σημαντικές, να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερα αποτελέσματα όχι μόνο να φέρουμε προ... τις δικαιοσύνης ε, αποτελεσματικά όσους ε, ε, έχουν προσδιοριστεί ότι εμπλέκονται, όσους έχει προσδιοριστεί ότι εμπλέκονται στο παρελθόν σε υποθέσεις διαφθοράς ο Γιαννουκόβιτς, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία που εκλάψαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τομέας πιστεύω είναι ένα πεδίο που κάνει καταπληκτική δουλειά η κοινωνία των πολιτών, χωρί όμω επαρκή υποστήριξη από εμά. Και όταν λέω εμά, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εμά ω κοινοβούλιο, δεδομένου ιδιαίτερα ότι τα περισσότερα ε, προϊόντα τη ε, διαφθόρα ε, βρίσκονται σε κάποια από τα δικά μα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε εντονότερα με την κοινωνία των πολιτών στην Ουκρανία, ώστε να αναλάβουν με την ευθύνη της καταπολέμησης διαφθορά, αλλά να μπορέσουν και να ανακτήσουν και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, τα οποία τόσο πολύ χρειάζεται η Ουκρανία. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Σόσνιες τώρα. Ja chciałem zaprotestować po raz kolejny przeciwko e, wszystkim. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θέλουμε όλες οι χώρες να υπογράψουν τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Δεν πρόκειται βέβαια για μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά ε, κάθε χώρα έχει, έχει τις αρμοδιότητές της. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποια χώρα να την υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Οπότε ε, διαμαρτύρομαι για το ότι μας παρουσιάζεται ως μια υποχρέωση. Η Πολωνία, για παράδειγμα, δεν έχει θεσπίσει αυτή την συμφωνία, δεν την έχει υπογράψει και είναι δικαίωμά τη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Να ζητήσω λοιπόν τον κύριο Γκάλερ να κλείσει τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι, για τα σχόλιά σας. Για τους περισσότερους πολίτες Ουκρανίας, πιστεύω, οι κοινωνικές συνθήκες είναι το ζήτημα που τους απασχολεί κατά κύριο λόγο στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφερθούμε εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα τώρα για τις άλλες ε, καταστάσεις, ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα όπως αναφέρθηκε. Αυτό είναι ένα θέμα όπου μαζί με τους πολίτες και τις πραγματικές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για ζητήματα όπως αναφέρατε και την αποκατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα χρήματα που ανήκουν στους πολίτες και στον εθνικό προϋπολογισμό. Όσον αφορά τη ζητήματα των μειονοτήτων, συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Σύνδεσης συζητήθηκαν εκτενώς. Εγώ θα κάνω και κάποια συζήτηση την επόμενη εβδομάδα για τις τροπολογίες σας και θα δούμε πώς, ε, τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Θα έχουμε και άλλη μια συνέντευξη σκιωδών και εκεί θα δούμε πώς, ε, ποιο, ποια είναι η διάθεση και οι απόψεις και θα συμπεριλάβουμε και την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της κυρίας Χάμς και του κυρίου Ροζάτη και με εσάς και αυτές θα ληφθούν υπόψη. Για το ζήτημα αυτό καθε αυτό πιστεύω θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η Ουκρανία να τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο που ισχύει ως νομοθεσία. Δεν πρέπει να δραματοποιούμε την κατάσταση, ούτε να λαμβάνουμε υπόψη εξτρεμιστικές απόψεις οποιασδήποτε ΜΚΟ ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας ως πολιτική ε, που ακολουθεί η Ουκρανία. Εξτρεμιστικές απόψεις ε, επί όλων των ζητημάτων υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Δεν μπορούμε να τις λαμβάνουμε υπόψη και να τις χρησιμοποιούμε ε, λέγοντας ότι αυτή την πολιτική ακολουθεί μια χώρα. Ό,τι αναφέρεται σε τέτοιο πλαίσιο δεν μας ενδιαφέρει ο εξτρεμισμός ουδέποτε και πουθενά δεν οδήγησε σε κάτι καλό. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις υποχρεώσεις που είναι υπαρκτές και να εκτιμήσουμε τι γίνεται με αυτό το νόμο και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. That concludes... Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Κλείνει έτσι η συζήτηση και για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα λάβει χώρα στις 12 Νοεμβρίου. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξή μας, εξαντλήσαμε και τους εαυτούς μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκούραση.